Υπάρχουν ορισμένες ανακοινώσεις από πλευράς του Προέδρου και μετά θα συνεχίσουμε με το κανονικό μας πρόγραμμα. Λόγω των τελευταίων δραματικών εξελίξεων στο Κίεβο, έχουν αποκτήσει μια νέα επικίνδυνη δυναμική. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς πως ξεκίνησαν πια τα πράγματα, αλλά και μετά από διαβουλεύσεις με την το εκπρόσωπο και τον επίτροπο Φούλε και τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μπροκ έφυγε και πάει στο Κίεβο για να είναι εκεί αύριο όπου θα συνέλθει η Βουλή για την ανάκληση των νόμων που ψηφίστηκαν στις 16 Ιανουαρίου, των αμφισβητούμενων νόμων. Ταυτόχρονα ο Επίτροπος Φούλε θα φτάσει σήμερα στο Κίεβο και η ε, ύπατη εκπρόσωπος θα πάει την Τετάρτη. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε το τι συμβαίνει στη νότια γειτονία μας και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο. Ξέρετε ότι θα έχουμε σύντομα συζητήσεις με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έτσι ώστε να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις στην Αίγυπτο. Και τέλος, και αυτό παραμένει σημαντικό γιατί έχουμε τον αξιότιμο πρέσβη της Τινησίας εδώ, να τον συγχαρώ για την υπερψήφιση και υπογραφή του νέου συντάγματος. Σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε η διαδικασία ε, θα ασχοληθεί με αυτό και ο κύριος Μπουκίκιο. Ζητά συγγνώμη ο κύριος Πάσκου από τον κύριο Μπουκίκιο. Λοιπόν, είναι πρόεδρος ο κύριος Μπουκίκιο της Επιτροπής της Βενετίας, τον καλωσορίζουμε και θα μας μιλήσει για την πολιτική μετάβαση στην ε, την Ισία, θα θίξει και τα της Τουρκίας και θα μας μιλήσει στο τέλος και για τη Λιβύη. Έχετε το λόγο κύριε Μποκίκιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας συγχαρώ καταρχάς γιατί επιλέξατε τη σημερινή μέρα για να συζητήσετε και τα της Ισίας. Χθες το βράδυ η, η συντακτική Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε με 200 ψήφους υπέρ 12 κατά και 4 αποχές το νέο σύνταγμα της Τινησίας. Ο πρόεδρος Ματσούκη πήρε το λόγο σήμερα το πρωί γιατί η τελετή για την υπογραφή έγινε σήμερα το πρωί της 11 είχα προσκληθεί ε, αλλά εγώ ε, προτίμησα να έρθω εδώ αλλά ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής της Βενετίας είναι εκεί ο κύριος Ματσούκη, ο πρόεδρος Ματσούκη αναφέρθηκε, ο πρωθυπουργός Ματσούκη αναφέρθηκε σε ένα σύμβολο για τη δημοκρατία και ο πρόεδρος Μπεντζαφάρ είπε ότι η σημερινή μέρα έχει τεράστιο βάρος, είναι μια πρωτοποριακή εμπειρία της Τινησίας, μια επιτυχία για την Τινησία και τη δημοκρατία. Συμφωνώ με αυτά τα οποία λοιπόν υπόθηκαν σήμερα στην Τίνιδα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τον Μάρτιο του 2012 έκανα την πρώτη επίσκεψή μου μετά από την Επανάσταση στην Τίνιδα, συνάντησα τις αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης και πολλές προσωπικότητες του νομικού κόσμου. Όλο τυχαίως ο κύριος Μπούζεκ, ο τέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δεν τον βλέπω εδώ σήμερα, θα ήθελα να τον χαιρετήσω, ήταν και αυτός εκεί και είχε προσφέρει ε, δείπνο, είχε καλέσει σε δείπνο το διπλωματικό σώμα των ευρωπαϊκών χωρών στην Τίνιδα και με είχε προσκαλέσει και μένα. Κατά τη διάρκεια του δείπνου έκανε μια, ένα, μια μικρή δημοσκόπηση και ζήτησε από τους συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν τις πιθανότητες εκδημοκρατισμού. Και δυστυχώς ξεκίνησε με μένα, ήμουν ο πρώτος στη σειρά τότε ήμουν έμπλεος αισιοδοξία μετά από τις πρώτες διαβουλεύσεις που είχα και είπα 7 στα 10 και ήμουν και ο μόνος που το είπα. Ε, ακολούθησαν οι πρέσβεις οι οποίες έδιναν από μία, από μία ψήφο ένα πόντο μέχρι πέντε πόντους ένιωσα άσχημα και πραγματικά ίσως υπερέβαλα από ενθουσιασμό. Σήμερα όμως τελικά είμαι ευτυχής γιατί η αισιοδοξία μου τεκμηριώθηκε και ευχαριστώ μέσω του πρέσβη τον λαό της Τινησίας. Τώρα λίγα λόγια για το ψήφισμα ε, για το σύνταγμα το οποίο υπεγράφει σήμερα. Καταρχάς η διαδικασία επεξεργασίας σύνταξη του νέου συντάγματος ε, ε, αν, ε, αναλήφθηκε από μια ειδική συντακτική λοιπόν που προτίμησε το λευκό χαρτί, να ξεκινήσει από λευκό χαρτί. Θα μπορούσε να εμπνευστεί από το πρόγραμμα που είχε προετοιμάσει η Επιτροπή του Προέδρου, του Μπεντζαφάρ, αλλά προτίμησε να ξεκινήσει από το μηδέν. Ισχυρή εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, και ε, πολύ ε, σε βάθος ε, νομική επεξεργασία θέσεων. Υπήρξε ένα άνοιγμα, όχι από την αρχή, αλλά που επιβεβαιώθηκε στην πορεία με την Επιτροπή της Βενετίας και με άλλα διεθνή φόρα, νομικά φόρα. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε πραγματικά σημαντικά βήματα. Το 2011 και το 2012 Κατά τη διάρκεια των περιοδικών συναντήσεων ανάμεσα στην Επιτροπή της Βενατίας ε, και τις έξι επιτροπές της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης μιλούσαμε ακόμα για τη Σαρία, για καταστολή, για ε, συμπληρωματικότητα άνδρα με γυναίκα, για εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ κτλ. Το 2013 και μετά από ε, πάρα πολύ μακρές συζητήσεις και σε ιδεολογικό επίπεδο και σε επίπεδο πραγματιστικό θα έλεγα οι έννοιες αυτές ευτυχώς χάθηκαν από το Σύνταγμα. Τον Ιούλιο του 2013 μετά από ένα αίτημα του Προέδρου Μπεντζαφάρ γνωμοδοτήσαμε σαν Επιτροπή Βενετίας για το σχέδιο έτσι όπως υπήρχε εκείνη την εποχή. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία θα έλεγα των συστάσεών μας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα το οποίο οδήγησε μετά τη σύνταξη του συντάγματος. Έχω την αίσθηση ότι το νέο σύνταγμα εσωτερικο, δηλαδή το, το ενσωμάτωσε ο λαός της Τινησίας. Δεν είναι μια απλή διακήρυξη θεμελιωδών δικαιωμάτων και οργάνωση των σχέσεων των κρατικών θεσμών. Πρέπει να είναι ικανό το κείμενο αυτό να εμπνεύσει ε, τον λαό της χώρας. Πρέπει να το αισθανθούν σαν δικό τους και όχι σαν ε, κάτι το οποίο επικρέμαται της χώρας τους αντικατοπτρίζει θα έλεγα το νέο κείμενο τις προσδοκίες και τις συμβιβαστικές λύσεις τις οποίες καταλήγει ο λαός της Τινησίας ελπίζω να υποστηρίξει στο μέλλον το σύνταγμά του. Για τον χρόνο τώρα, ο οποίος απαιτήθηκε για αυτή την πρωτοβουλία, τρία χρόνια, είναι άραγε υπερβολικό. Ενθυμούμε γιατί όπως ξέρετε <clears throat> είχαν υπάρξει κάποιες προθεσμίες που είχαν καθοριστεί και οι οποίες ε, κάθε φορά τις ξεπερνούσαν. Αλλά κάθε φορά έλεγα ότι πράγματι αυτό το οποίο κάνουμε εδώ είναι ένα σύνταγμα. Πρέπει όμως να είναι ένα καλό σύνταγμα. Δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί. Δεν πρέπει φυσικά να κολλησιεργούμε, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι με σωστό ρυθμό. Τρία χρόνια ίσως να είναι λίγο μεγάλος ο χρόνος, αλλά ήταν απαραίτητος. Υπήρξαν και άλλοι λόγοι. Καταρχάς η συντακτική εθνοσυνέλευση δεν είχε μόνο αυτή τη δουλειά, είχε και τακτικές νομοθετικές αρμοδιότητες, νομοθετούσε πάνω σε πάρα πολλά θέματα. Η συντακτική αυτή εθνοσυνέλευση χρειάστηκε χρόνο για τον καθορισμό και του εσωτερικού της κανονισμού του εσωτερικού της κανονισμού λοιπόν και κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή τη συνταγματική έστω και με κάποια καθυστέρηση. Υπήρξαν και ε, πολιτικά προβλήματα, ακόμα και τραγωδίες, απόπειρες, ε, δολοφονίες, αλλά όλα αυτά επιβράδυναν τη διαδικασία. Τώρα, για το περιεχόμενο ε, του συντάγματος, ε, μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχαν τροποποιήσεις, οπότε εδώ ίσως διακινδυνεύω λίγο γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς την τελική διατύπωση. Παρόλα αυτά, ε, σε επίπεδο γενικών γραμμών πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για το περιεχόμενο. Καταρχάς, μιλάμε για τον καθαρά δημοκρατικό πολιτικό χαρακτήρα του κράτους που βασίζεται στην ιδιότητα του πολίτη, στην λαϊκή κυριαρχία και το δίκαιο των πολιτών. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία της Τινησίας. Αυτή η διατύπωση είναι πολύ καλύτερη από το να πούμε ότι το Ισλάμ είναι κρατική θρησκεία ή θρησκεία του κράτους. Στην ουσία χρησιμοποιήθηκε εκ νέου η διατύπωση του Μπουργκιμπά του 76 που είχε σαν στόχο να ευνοήσει το λαϊκό κράτος και νομίζω ότι ήταν ένα καλό βήμα. Σε επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπάρχει σημαντική πρόοδος. Τα περισσότερα αναγνωρισμένα θεμελιώδη δικαιώματα από τις διεθνείς συμβάσεις υπάρχουν. Πολιτικές ελευθερίες, διαδήλωσης, συνέβρεσης κτλ. Όπως το προβλέπει και η Επιτροπή της Βενετίας. Λέγεται ότι κάθε περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η ισότητα σε επίπεδο δικαιωμάτων είναι, ανήκει και στους άνδρες και στις γυναίκες χωρίς καμία διάκριση. Προβλέπεται επίσης ότι το κράτος κάνει κάθε προσπάθεια για την εγγύηση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στα εκλεγμένα σώματα σε όλα τα επίπεδα. Η ισότητα των ευκαιριών επίσης έχει γίνει αντικείμενο εγγύησης. Υπάρχει μια ρήτρα σχετικά περιοριστική, δεν ξέρω αν έχει μείνει. Ε, υπάρχει και ένα σημείο αρνητικό αλλά δεν είναι καθοριστικό. Η ρήτρα αυτή λέει ότι υπάρχει ε, ε, ε, ισότητα, ευκαιριών για να αναλάβει το κάθε φύλλο τις διαφορετικές του ευθύνες, λέει το κείμενο. Η ελευθερία πίστης είναι κάτι το οποίο γίνεται αντικείμενο εγγύηση σε επίπεδο κρατικού καθήκοντος περισσότερο και όχι σαν ατομικό δικαίωμα το πολιτικό καθεστώς είναι ημιπροεδρικό. Ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα σε δύο γύρους, με δύο γύρους για μία πενταετία όπως και η Εθνοσυνέλευση. Αυτό είναι καλό γιατί αποτρέπει ε, πιθανές ε, ε, αυταρχικές τάσεις. Ο Πρωθυπουργό ορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών και είναι υπόλογος προς το Κοινοβούλιο. Οι εξουσίες του Προέδρου είναι σημαντικές, είναι υπεύθυνο για τις εξωτερικές υποθέσεις, για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια και μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες συγκρούσεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο. Όμως υπήρχε και υπάρχει ε, ε, μια, ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο προβλέπεται το οποίο οφείλει να είναι ουδέτερο και δίκαιο και πιθανώς αν υπάρχουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων θα κρίνονται από το ανώτατο αυτό συνταγματικό δικαστήριο. Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας είναι κάτι που αμφισβητήθηκε στην Ισία. Το σχέδιο συντάγματος καθορίζει τις αρχές της κυριαρχίας της δικαστικής και του δικαστή του σεβασμού των αρμοδιοτήτων του και την μη δυνατότητα μετακίνησής του. Δημιουργείται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα η σύστασή του, με μια μεγάλη πλειοψηφία δικαστών. Βέβαια αυτό δεν αρκεί. Ένα από τους βασικούς στόχους της συντακτικής συνέλευσης ή και του νέου κοινοβουλίου μετά τις επόμενες εκλογές είναι μια μεταρρύθμιση σε βάθος του δικαστικού συστήματος της χώρας. Λοιπόν, το Σύνταγμα θα τεθεί προοδευτικά σταδιακά σε λειτουργία. Εν τω μεταξύ η συντακτική θα συνεχίσει να νομοθετεί και αυτό μέχρι τις επόμενες εκλογές. Στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμα, θα οργανωθούν τέσσερις μήνες μετά από τη θέση σε ισχύ του νέου Συντάγματος. Όμως νομίζω ότι ε, θα οργανωθούν τελικά στις αρχές του φθινοπόρου. Αυτό είναι καλό. Το κόμμα έναντα και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Χανούτσι, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει εκλογές ανάμεσα στο μήνα Ιούνιο και το μήνα Οκτώβριο. Νομίζω ότι και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα θα συμφωνήσουν με το κόμμα Εναντά, οπότε ελπίζουμε οι εκλογές ε, να γίνουν ε, σύντομα, φέτος. Ο εκλογικός νόμος ε, θα, θα συνταχθεί τις επόμενες έξι εβδομάδες. Ίσως αυτό να μην ακούγεται πολύ ρεαλιστικό, αλλά είναι μια προσπάθεια, θα γίνει μια προσπάθεια, θα πάνε γρήγορα τα πράγματα. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ήδη συνεκλήθη, εννέα μέλη έχουν ήδη οριστεί. Ο Μπεντζαφάρ έλεγε στο τέλος της ομιλίας του εδώ και δύο ώρες ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Θα πρέπει να επιβεβαιωθούν οι δημοκρατικές αρχές. Η προτεραιότητα είναι πλέον η οικονομία και το άνοιγμα των αγορών. Θα πρέπει δηλαδή να οικοδομηθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί σε όλα τα επίπεδα και στην οικονομία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν πρόεδρε σήμερα ότι εμείς πιστεύουμε και στηρίζουμε το τινησιακό πρότυπο και ελπίζουμε να εξαχθεί και στις υπόλοιπες χώρες περιοχής. Oui, je peux, je peux, να συνεχίσω. Μια και είμαστε στην ε, ευρύτερη περιοχή, να μιλήσω για την ε, Λιβύη. Ήμουνα 7 με 9 Ιανουαρίου στην ε, Τρίπολη και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. το Κογκρέσο, δηλαδή η Εθνοσυνέλευση της Λιβύης δεν έχει πια την εμπιστοσύνη του λαού, ο Πρωθυπουργό Αρσεϊντάν δεν χαίρει τη εμπιστοσύνη του λαού της Λιβύης και ενό σημαντικού τμήματο τη Βουλή της Λιβύης, οπότε η κατάσταση είναι ασταθής. Κατά την επίσκεψή μου εκεί και στη συνάντηση με βουλευτές συζητήσαμε τρία κυρίω θέματα. Το πρώτο ήταν κατά πόσο το Κογκρέσο, η Βουλή της Λιβύης θα πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία του 7 Φεβρουαρίου, κάτι που δεν φαινόταν σε κανένα συνταγματικό κείμενο, ούτε στην συνταγματική διακήρυξη, η συντακτική διακήρυξη της, του Κογκρέσου. Υπάρχουν προθεσμίες για τα διάφορα καθήκοντα του Κογκρέσου, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται ότι θα πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία του 7 Φεβρουαρίου το Κογκρέσο της Λιβύης. Οπότε μπορεί να συνεχίσει. Βέβαια υπάρχει μια πρόταση μορφής ε, κατά του Πρωθυπουργού. Μέχρι στιγμής όμως καμία πολιτική δύναμη δεν συγκέντρωσε τις 120 ε, απαραίτητες ψήφους για να ευοδοθεί αυτή η πρόταση μορφής και μιλήσαμε και για την συντακτική συνέλευση, ε, την σύσταση μιας ε, συντακτικής επιτροπής γιατί η επιτροπή αυτή θα πρέπει να έχει 60 μέλη, η εκλογική διαδικασία για τη σύστασή της έχει ολοκληρωθεί και αν δεν δημιουργηθούν προσκόμματα ή περαιτέρω αστάθεια, θα πρέπει στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου να συγκροτηθεί, να συνεδριάσει αυτή η περαιτερω ασταθεια θα πρεπει στα δευτερο μισο Αυτή η εκλεγμένη Επιτροπή, που είναι πολύ πιο λιγομελής από την ε, συντακτική συνέλευση της ε, την ε, δεν θα έχει νομοθετικές αρμοδιότητες, θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το Σύνταγμα και θα μπορέσει να ξεκινήσει τις εργασίες της. Εμείς είπαμε ότι είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε αυτή την Επιτροπή. Υπάρχουν προβλήματα με τις μειονότητες, το ΑΡΕΓΑ, ΝΑΖΙΚ. Ιδιαίτερα οι ΑΝΑΖΙΚ ζήτησαν να συμπεριληφθούν στο Σύνταγμα να γνωριστεί ως επίσημη η γλώσσα τους, η μητρική τους γλώσσα. Αυτά τα θέματα ελπίζουμε ότι θα διαθετηθούν στο μέλλον γιατί είναι μεν σημαντική η γλώσσα αλλά υπάρχουν άλλα δικαιώματα των μειονοτήτων που είναι ακόμη πιο σημαντικά. Πρόσβαση στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, δυνατότητα να έχουν δικούς τους ε, ραδιοτηλεπτικούς σταθμούς. Αυτό είπα λοιπόν στη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Αναζίγκο, ότι εμεί θα είμαστε οι θεματοφύλακε των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Λιβύη. Ευελπιστούμε ότι η κατάσταση στη Λιβύη θα εξελιχθεί θετικά. Για την Τουρκία και εδώ έχω μια χαρμόσυνη σχετικά είδηση, γιατί είχαμε όλοι ανησυχήσει τα μάλα από την κατεύθυνση που ε, φάνηκε να παίρνει η κυβέρνηση με τον νόμο αυτό για τη μεταρρύθμιση του ΥΠΑ του Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων που παλιδρομούσε αισθητά σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του 2010 και το συνταγματικό πακέτο. Εγώ προσωπικά και ολόκληρη σύσσωμη Επιτροπή της Βενετίας ε, εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο και μάλιστα ε, είχαμε συστήσει και ένα συμβούλιο ε, των δικαστών που περιλάμβανε και τους εισαγγελείς και χωρίς είναι τέλεια αυτή η πρόταση βαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα τότε και μέχρι σχετικά πρόσφατα ο Υπουργό Δικαιοσύνη Σαντουλά Έργκιν ουδέποτε δεν προέδρευσε στο Συμβούλιο αυτό παρά μόνο μία φορά, οπότε συστηματικά απήχε. Ήταν μάλλον τυπική αυτή η προεδρία δηλαδή. Και η προτινόμενη μεταρρύθμιση ήταν ακόμη πιο φιλόδοξη. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη ε, θα είχε πολύ περισσότερε εξουσίε και όχι μόνο τυπικέ αλλά και ουσιαστικέ. Ο κύριο Τσίτσεκ, όπω ξέρετε, ο πρόεδρο τη ε, Τουρκική Εθνοσυνέλευση, δήλωσε πριν από δύο μέρε ότι η συζήτηση για τα θέματα αυτά, για το είπα Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων, ε, έχει διακοπεί και μάλιστα θα γίνει συζήτηση με τις ε, δυνάμεις αντιπολίτευσης προκειμένου να θεσπιστούν πιο μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Προς το παρόν όμως απετράπει ο κίνδυνος. Ε, αυτά και είμαι στη διάθεσή σας κύριε Πρόεδρε για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Έχουμε μια πληθώρα πολύ πρόσφατων πληροφοριών και μια και πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας στις 4 ακριβώς. Θα ήθελα να θερμοπαρακαλέσω τους εγγεγραμμένους μας αγορητές να περιοριστούν στο 1,5 λεπτό ο καθένας. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής της Βενετίας, σας ευχαριστούμε θερμά για το έργο της Επιτροπής σας, όχι μόνο στις χώρες της ε, Αραβικής Άνοιξης, αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Ουκρανία Εκεί ξέρω ότι συμβάλλατε ώστε... Παρακαλώ να σταματήσει το χρονόμερο, το χρονόμετρό μου κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για το έργο της Επιτροπής σας, όχι μόνο στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, αλλά και σε άλλες χώρες όπως την Ουκρανία, που έχουμε προβλήματα και διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης όπως είπατε πολύ σωστά, το θέμα του συντάγματος της θυνησίας, παρά τις όλη όλης διαδικασίας κατέληξε σε αίσιο πέρας και είπατε κι εσείς ότι είναι πιθανό και σχεδόν βέβαιο ότι οι εκλογές θα γίνουν φέτος. Ποιος είναι ο δικός χάρτης αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Πώς θα διεξαχθούν. Έχετε κάποιες ιδέες για τις για την πιθανή ημερομηνία ή το Σύνταγμα προβλέπει κάποιο χρονικό ορίζοντα για τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών. Τώρα, για τη Λιβύη που είπατε, δεν ξέρω αν είναι στο δικείμενο της συζήτηση, αλλά θα ήθελα να μου κάνετε μια αξιολόγηση με την πλούσια πείρα που έχετε ως πρόεδρος της Επιτροπής Βενετίας για το πρόσφατο συνταγματικό κείμενο που εγκρίθηκε στην Αίγυπτο. Τι γνώμη έχετε για το νέο σύνταγμα της Αιγύπτου. Θεωρείτε ότι βελτιώνει την το προηγούμενο σύνταγμα. Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε μια έγκριτη και αντικειμενική αξιολόγηση από εσά. Γιατί δεδομένων των εξελίξεων και των γεγονότων στην Αίγυπτο, μια τέτοια αξιολόγηση ήταν πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως ε, για την παρουσία σας ε, κύριε Πουκίκιο και για τις ε, καλές ειδήσει που μας φέρατε. Θα ήθελα μερικές πληροφορίες για ορισμένα στοιχεία του, συντάγματος, του νέου συντάγματος της Τινησίας. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τις εξελίξεις και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η διατύπωση για το ρόλο της Σαρίας ε, του Ισλαμικού νόμου. Γιατί όχι μόνο στην Τινησία αλλά και οι γειτονικέ χώρες μας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη διατύπωση που βρέθηκε, ιδιαίτερα στο Σύνταγμα της Τινησίας. Ποια ήταν η λύση που επιλέχθηκε. Επίσης, θα ήθελα να μάθω αν ενισχύθηκε η ανεξαρτησία της, του δικαστικού κλάδου, της δικαιοσύνης. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Διάβασα ότι σε ό,τι αφορά το σεβασμό των διεθνών συνθήκων και συμβάσεων, ίσως η διατύπωση του συντάγματος δεν είναι και πολύ καλή. Λέει, ε, στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν στο σύνταγμα οι διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Αν ισχύει αυτό, θα δημιουργούνται ένα πολύ κακό προηγούμενο και δεδομένη της ε, σχετικής νομολογίας που υπάρχει. Πάντως ε, ήταν σημαντικό το γεγονός ότι εγκρίθηκε τελικά το Σύνταγμα στην Τινησία. Για τη Λιβύη είχα πάει τον Νοέμβριο και όντως η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ και για την Αίγυπτο αλλά και για την Τουρκία πέραν ε, της κατάργησης ή της ε, μη αυτού του απειλητικού αυτού νόμου. Τι γίνεται με τις απειλές που εξαπειλήθηκαν κατά, το, δικαστών και του δικαστικού κλάδου γενικώ. Ο κύριος Νταφ. Καλησπέρα σας. Πρόεδρε, χάρηκα βεβαίως όταν άκουσα ότι η νομοθετική διαδικασία στην Τουρκία έχει ε, σταματήσει για αυτό το νέο νόμο. για τους δικαστές ε, και τους ε, εισαγγελείς, αλλά δεν θα πρέπει να γελιόμαστε, ούτε εμείς, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε κανένας άλλος. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι γνωρίζει βαθιά κρίση ε, του κράτους αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Έχει φτάσει στα πρόθυρα της παραβίασης των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Διότι δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την ίδια την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Πώς είναι δυνατόν αυτό χωρίς παραβίαση λέγω των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Ο Πρωθυπουργός Ερντοάν την περασμένη εβδομάδα ήταν στις Βρυξέλλες και εμφανίστηκε έτσι με κάποιο βελτιωμένο λεξιλόγιο, ε, με μια πιο μετριοπαθή, συγκρατημένη ε, ρητορική και διατύπωση στα λεγόμενά του σε σχέση με το παρελθόν. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια στιγμή απέλυε ή έπαβε δικαστές και ε, εισαγγελείς στην Τουρκία. Σε ευρύτατη όσο και ανισχυτική κλίμακα. Ερωτώ λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος ε, Τσίτσεκ είναι σοβαρά διατεθειμένος να συνεργαστεί με την Επιτροπή της Βενετίας ε, με σκοπό τη βελτίωση του σχεδίου ε, του σχετικού νόμου. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεναράμπ Ατού. Euh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ όπως και οι συνάδελφοί μου να χαιρετήσω τους την για ε, το σύνταγμα αυτό και να του συγχαρώ. Ήταν πραγματικά δύσκολη αυτή η υπόθεση αλλά στέφθηκε με επιτυχία και θέλω να συγχαρώ το λαϊνό της Τινησίας για την ευφυΐα και το θάρρος. Θέλω να αναφερθώ στις χώρες Μακρέπ ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα το πρώτον. Στο νέο Σύνταγμα της Τινησία γίνεται λόγος για το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Διότι έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το διακύβευμα. Αν δει κανείς πώς τα ακραία κόμματα χρησιμοποιούν ή ε, εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά ζητήματα για να κατακτήσουν την εξουσία, τα δημοκρατικά κόμματα δεν μπορούν να τα αγνοούν. Ε, είπατε ότι ο κύριος Μπεντζαφάρ αναφέρθηκε στην ανάγκη διάνοιξης των αγορών. Μήπως κινδυνεύει να πέσει στο ίδιο σφάλμα η Ισία με την Ευρώπη, δηλαδή να αρχίσει μια ε, φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, γιατί με ανισχύει αρκετά αυτό το θέμα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Ένωσης του Μαγκρέμπ. Ξέρω ότι ο κύριος Μαρζουκή ήθελε να ε, ανακοινήσει αυτό το θέμα, δεν το κατάφερε γιατί βεβαίως η Αλγερία και το Μαρόκο είναι οι δύο πρωταγωνιστές και για την Αλγερία το 2014 θα είναι κρίσιμη στιγμή με προεδρικές εκλογές. Εσείς πώς αναλύετε την κατάσταση της Αλγερίας, την εξουσία στην Αλγερία και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης εκεί στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκάλερ που είναι πρώην επικεφαλής των παρατηρητών στην ε, την Ισία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και υπό την ιδιότητα αυτή ακριβώς θα ήθελα να τονίσω πόσο χαρούμενος είμαι και με πόσο μεγάλη ανακούφιση καλωσορίζω αυτό το αίσιο αποτέλεσμα. Παραδέχομαι ότι με τη σειρά των μήνων είχα την ε, εντύπωση ε, όλους αυτούς τους μήνες ότι ε, θα μπορούσε και να εκτροχιαστεί όλη η υπόθεση. Τελικά ε, πριτάνευσε και κυριάρχησε η λογική και το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα είναι καλό για την Τινησία και το λαό της και μπορούμε να τους συγχαρούμε και πρέπει να τους συγχαρούμε. Αλλά θα πρέπει να συγχαρούμε λίγο και τον εαυτό μας, γιατί και η Ευρώπη έκανε καλές προτάσεις, είτε πρόκειται για την Επιτροπή της Βενετίας που διαδραμάτισε ένα εξαιρετικό ρόλο και σας ευχαριστώ για αυτό, αλλά και για όλες τις άλλες δραστηριότητες που έχετε εκεί σε αυτό το τομέα. Αλλά είχαμε και μια ε, επιτροπή συντονισμού, θέλετε, κομιτέντε πιλοτάζ, που ε, παρακολουθούσε όλη αυτή τη διαδικασία και οικονομικά όλη η κοινότητα των δωρητών. Ήταν κρίσιμο και αυτό να ε, γίνει δουλειά και με προτάσεις και από αυτή τη σκοπιά. Έρχομαι τώρα να ρωτήσω το εξής επειδή με ταχύς ρυθμούς τώρα πλησιάζουν οι εκλογές, έχετε την αίσθηση ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ε, έχει προετοιμαστεί σωστά και μπορεί να τηρηθεί το προβλεφθέν χρονοδιάγραμμα και υπάρχει πολιτική συνένεση ε, σε κόμματα ε, κοινοβουλευτικά που δεν συμμετείχαν σε αυτή τη ε, συντακτική συνέλευση. Πώ το κόμμα είναι Τούνη, πώ το σκέφτεστε αυτό, πώ το βλέπετε. Κυρία Ντεκεζέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μποκίκιο, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είναι γεγονό ότι τα νέα που μας έρχονται από την, την Ισία είναι πολύ αισιόδοξα σε σχέση με τη χώρα αυτή που ήταν η πρώτη που ξεσηκώθηκε στην ε, Αραβική Άνοιξη. Ξέρω ότι δεν θα είχαν ε, στοιχηματίσει πολύ, δεν θα είχαν ποντάρει σε αυτή την επιτυχία. Εγώ θυμάμαι ότι είχα προσκληθεί στη Τινησία να συμμετάσχω σε συνεδριάσεις της συντακτικής συνέλευσης. Ήταν πάρα πολύ ζωντανές οι συζητήσεις και ε, μέσα σε ένα επαναστατικό πνεύμα είτε ήταν ε, εκπρόσωποι των κομμάτων εναχτά, τα κατόλοι, άλλο. Έχω να ρωτήσω το εξή Τι γίνεται με τις χώρες που δεν κατάφεραν να επιτύχουν αυτή την εξέλιξη. Όταν ο πρόεδρος Μόρση στην Αίγυπτο ε, είχε αρχίσει αυτή τη συντακτική του προσπάθεια, ε, είδαμε ότι δεν ανταποκρινόταν στα δημοκρατικά πρότυπα. Και τότε είχα ζητήσει από τον Επίτροπο Φίλε και μετά από συζήτηση με ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κάιρο, ε, Είχα λοιπόν ρωτήσει τον κύριο Φίλε μήπως θα μπορούσαμε να στείλουμε όχι ακριβώς προειδοποίηση αλλά ένα μήνυμα. Προσοχή, να κρούσουμε ένα κόδωνα κινδύνου. Και τότε φάνηκε δύσκολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, παρέμβει σε μια συντακτική ε, συνέλευση, μια διαδικασία ε, που ήταν ζήτημα του ίδιου του λαού. Όταν έχουμε τέτοιες όμως εξελίξεις, τρευλές, όπως στην Αίγυπτο, τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα, γιατί δεν είναι σε σωστό δρόμο η ε, Αίγυπτος υπάρχουν νεκροί. Είναι ένα τρελό τρένο το οποίο έχει εκτροχιαστεί. Ο κύριος Κύριλοφ, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η ερώτησή μου ίσως και να έχει ήδη τεθεί. Θα ήθελα πάντως να επανέλθω στην Τουρκία. Θα ήθελα τη γνώμη σας κύριε Μπουκίκιο γύρω από την ισχυρότατη επιρροή του κινήματος Φέτβα Γκιούλεν. Στο παρελθόν υπήρχε μια κάποια όχι ιδιαίτερα σταθερή ε, αλλά συνένεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο κίνημα σχετικά με τον ρόλο του καθενός. Κάτι τέτοιο λειτουργήσε θετικά. Πώς βλέπετε όμως από εδώ και πέρα την κατάσταση, ιδιαίτερα μετά από τις τελευταίες ε, εξελίξεις που φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια ε, αναδιάταξη των θέσεων και υπάρχουν και πολιτικές κινήσεις εις βάρος του συγκεκριμένου κινήματος. Θα ήθελα επίσης να πω στον κύριο Μπουκίκιο σχετικά με το ρόλο της ε, Επιτροπής της Βενετίας. Εγώ ήμουνα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και πράγματι νομίζω ότι ε, δίδεται μια καλύτερη ορατότητα και μια καλύτερη και ισχυρότερη εικόνα ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κάτι το οποίο θα βοηθήσει να πετύχετε τα, τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμείτε. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για τις ερωτήσεις σας. Θα τις ε, ομαδοποιήσω πριν τις απαντήσω. Για την εκλογική διαδικασία. Υπάρχει στο νέο σύνταγμα το άρθρο 143 που προβλέπει ότι οι εκλογές θα πρέπει να οργανωθούν τέσσερις μήνες μετά από τη θέση σε ισχύ του συνταγματικού χάρτη, από σήμερα δηλαδή. Ή μάλλον λέει το άρθρο δεν μπορούν να γίνουν οι εκλογές πριν περάσουν τέσσερις μήνες. Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε τέσσερις μήνες. Αν μείνουμε σε αυτήν την όθηση τη συνενετική η οποία υπήρχε και στην αίσθηση εθνικής ενότητας των πολιτικών δυνάμεων της χώρας που έδειξαν μια τέτοια ευθύνη, νομίζω ότι μπορεί να το πετύχουν όπως ακριβώς προβλέπεται μέχρι το φθινόπωρο ή πριν το τέλος του χρόνου, εν περιπτώσει. Αυτό έχει σημασία έχει σημασία γιατί θα είναι αν θέλετε το τελευταίο βήμα για το πρώτο επίπεδο σταθεροποίησης της χώρας, δηλαδή νέες εκλογές, νέος πρόεδρος, νέο σύνταγμα. Κύριε Γκάλερ, το όργανο στο οποίο αναφερθήκατε λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στις πρώτες εκλογές της, στην ε, την Ισία και θα κάνει την ίδια και εξαιρετική δουλειά και τώρα. Απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις έτσι ώστε να οργανωθεί σωστά η εκλογική διαδικασία και να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά σχέδια για τον εκλογικό νόμο, κάποια προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών που είναι ιδιαίτερο θετικά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έξι εβδομάδες επαρκούν σαν χρόνος έτσι ώστε να κλείσει το νέο κείμενο. Πάντως νομίζω ότι ο νέος εκλογικός νόμος θα γεννηθεί στην την Ισία συντομότατα. Αναφερθήκατε στη Σαρία. Η Σαρία δεν υπάρχει στο νέο σύνταγμα. Καταρχάς δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε τη Σαρία. Ε, η Σαρία θα πρέπει να ερμηνευθεί φυσικά από τους θρησκευτικού ηγέπτες και στην Αίγυπτο η ερμηνεία που δίδεται είναι αρκετά φιλελεύθερη. Οι Τινήσοι όμως πήγαν και πέραν αυτού. Εάν ήθελαν να συμπεριλάβουν την Σαρία σαν πηγή δικαίου, αυτό δεν ε, λειτουργήσε. La justice. La justice, ε, Για τη δικαιοσύνη τώρα. Όπως είπα, το θέμα της δικαιοσύνης είναι πρόβλημα στην Τινησία. Υπάρχουν τα θεμέλια στο νέο σύνταγμα, αλλά η μεταρρύθμιση του δικαστικού είναι προτεραιότητα. Ιδιαίτερα σχετικά με την εκπαίδευση των δικαστών, τους εφαρμοστικούς νόμους, εφαρμοστικές διατάξεις μάλλον κτλ. Είναι ένα θέμα στο οποίο οι νέες αρχές και ήδη και η συντακτική όσο έχει την ομοθετική εξουσία πρέπει να δώσουν ιδιαίτερο βάρος. Για την Ένωση του Μαγκρέμπ, συγγνώμη αγαπητή μου κυρία, εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά αυτήν την ε, μορφή ε, σύνδεσης που κάνατε και δεν θα απαντήσω σε αυτή. Όταν ο Μπεντζαφάρ έλεγε ότι πρέπει να ανοίξουν οι αγορές, αυτό που ήθελε να πει είναι ότι θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε να επιστρέψουν οι επενδύσεις που φύγαν μετά την Επανάσταση. Ξέρετε, υπέφερα από τρία δεινά η την Ισία, την ίδια την Επανάσταση, το μισό εκατομμύριο Λιβύους πρόσφυγες, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτός και την οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Μην το ξεχνάτε αυτό, ήταν σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για μας αλλά και για τους Τινήσιους. Πολλές επιχειρήσεις που είχαν μετακινηθεί στην Τινησία επέστρεψαν στην Ευρώπη. Ελπίζω τώρα ότι στα πλαίσια της νέας σταθερότητας θα έλεγα αυτοί οι επενδυτές θα επενδύσουν εκ νέου στην Τινησία και θα καλύψουν λίγο την ανεργία η οποία χαίνει στην περιοχή. Για την Αίγυπτο τώρα. Η Επιτροπή της Βενετίας δεν έχει ασχοληθεί ε, με το νέο σύνταγμα το οποίο υιοθετήθηκε με το δημοψήφισμα της Αιγύπτου. Είχαμε κάποιες επαφές, το σύνταγμα αυτό από ό,τι φαίνεται δεν είναι ικανοποιητικό Υπάρχουν κάποια βήματα προοδού σε σχέση με τα βήματα που είχαν γίνει στο Σύνταγμα που είχε ψηφίσει η Προεδρία Μόρση. Πάντως ε, πολλές πολιτικές δυνάμεις τότε δεν είχαν πάρει μέρος στην επεξεργασία α, του νέου συντάγματο. Δυστυχώ το ίδιο έγινε και τώρα. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι δεν θέλησαν να συνεργαστούν με την λεγόμενη ομάδα των πεντήκοντα που επεξεργάστηκε το νέο σύνταγμα. Υπάρχουν πολλά που μένει να γίνουν λοιπόν. Τι μπορεί να γίνει τώρα με την διεθνή κοινότητα, τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα. Δρά η διεθνής κοινότητα. Το είδαμε αυτό και στην Ουκρανία και στην Τουρκία, το είδαμε και στην Τινησία και στη Λιβύη είναι παρούσα. Και στην Αίγυπτο. Μερικές φορές η διεθνής κοινότης δρά με μεγάλο δυναμισμό, άλλες φορές με μικρότερο δυναμισμό, της ελείπει μια κάποια ευελιξία. Εγώ βλέπω σε περιπτώσεις όπου στο Νότιο Κάφχασο, σαν παράδειγμα, που έπρεπε να υπάρχει μια πιο ισχυρή αντίδραση, Δυστυχώς οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας υπαγορεύονται ίσως από άλλα συμφέροντα. Όμως στην Αίγυπτο η διεθνής κοινότης ε, είχε κάπως μπλοκαριστεί γιατί αμέσως μετά την Επανάσταση ο Αιγυπτιακός πληθυσμός ήταν κατά γενικότερα των παρεμβάσεων του διεθνούς παράγοντα και ήταν δύσκολη η δράση της. Πάντως μπορώ να πω ότι χάρη στη δράση ε, του ειδικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κυρίου Λαμπρινίδη που πήγε στην Αίγυπτο και έπεισε τον πρόεδρο Μόρση να ζητήσει την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας για τις δημόσιες διαδηλώσεις. Το είχε πετύχει ο κύριος Λαμπρινίδης αυτός. Συνεργαστήκαμε με το γραφείο του Μόρση λοιπόν, αλλά δυστυχώς πριν ψηφιστεί ο νόμος σύμφωνα με τις δικές μας προτάσεις είχε ανατραπεί ο πρόεδρος Μόρση και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Αν μας φωνάξουν θα είμαστε έτοιμοι. Δεν αυτοεπιβάλλεται η Επιτροπή της Βενετίας, προσβλέπουμε στους φίλους και εταίρους την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να μοιραστούν μαζί μας όχι τα δικά μας μαθήματα αλλά τις κοινέ εμπειρίες τις οποίες τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ζήσει στην Ευρώπη μετά από την πτώση του τείχους. Τώρα για τα της Τουρκίας. Η κατάσταση στην Τουρκία είναι θα έλεγα σοβαρή, κρίσιμη. Ε, ίσως εσείς να είστε πιο αισιόδοξο από μένα για την Τουρκία. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μια κρίση στην παρούσα φάση συγκυριακή. Περιμένω τις επόμενες εκλογές και θα ξεκινήσουμε ήδη από τις δημοτικές εκλογές για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σύσταση της πολιτικής σκηνής. Υπάρχουν όμως κάποιες ενδείξεις για αρνητικές εξελίξεις σε πολλαπλές περιπτώσεις και σε κοινωνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο και σε δικαστικό νομικό επίπεδο. Όλες οι προσπάθειες τις οποίες από κοινού κάναμε για την συνταγματική αναθεώρηση δεν ολοκληρώθηκαν, έχουν τεθεί στον καταψύκτη προς το παρόν. Αυτό που είπε η κυβέρνηση πρόσφατα, ότι θα συζητήσουν με την αντιπολίτευση για να υπάρξει μια μεταρρύθμιση σε μεγαλύτερο βάθος μεταξύ μας, νομίζω ήταν ένα άλοθη της κυβέρνησης για να μην δείξει ότι παναχωρούσε Και μιας και μιλάμε για το ρόλο της διεθνούς κοινότητας θα ήθελα να πω ότι η παρέμβασή μας επηρέασε θετικά. Υπήρξαν δηλώσεις του κυρίου Γιάγκλαν, του Γενικού Γραμματέα του Συμβολίου της Ευρώπης, υπήρξαν δηλώσεις του Βαν Ρόμπαϊ, του Μπαρόζο και κυρίως να μην ξεχνάμε και σε εθνικό επίπεδο υπήρξε μια κινητοποίηση πολύ σημαντική. Ακόμα και ο πρόεδρος Αμπτουλαγιούλ είπε και διαβάζω το τι είπε ότι η συμβατότητα με το λεγόμενο άμεσο δημοκρατικό επίπεδο είναι κρίσιμη για τις χώρες μας όπως υποδεικνύεται από τα διεθνή όργανα όπως η Επιτροπή της Βενετίας κάτι το οποίο θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα δικά μας νομικά συστήματα. Ε, λειτουργεί διαιτητικά ο πρόεδρος, δεν έχει τις εξουσίες, δεν είναι πρωθυπουργό, αλλά υπάρχουν δυνάμεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, ακόμα και στο εσωτερικό του κυβερνητικού κόμματος, που ε, τίνουν να πιέζουν προς τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και σε διεθνές επίπεδο. Και ο συνάδελφός μας, ο κύριος Τσουρασούλου, ο οποίος είναι μέλος ε, της Επιτροπής μας, έχει διατελέσει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που γνωρίζει ποια είναι τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά στάνταρτς. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε σωστά μαζί του. Μη είμαι βέβαιος ότι δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας, αλλά ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και θα σταματήσω εδώ. Η κυρία Μπεναμπάρα Του θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Κύριε Μπουκίκιο, δεν απαντήσετε στην ερώτηση για την ε, κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Αναφέρθηκε τίποτα στις διαπραγματεύσεις και υπάρχει κάτι σχετικό στο Σύνταγμα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Συγγνώμη κυρία Μπεναμπάρα του. Όπως είπα, η πλειοψηφία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Ε, υπάρχει εγγύηση και κατοχύρωση του δικαιώματος του συνδικαλίζεστε. Το δικαίωμα στην εργασία επίσης τη χάνει εγγύησης. Και μάλιστα ε, αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά κοινωνικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα. Ευχαριστώ. We also have a request. Και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε το λόγο παρακαλώ εν συντομία. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το λαό της Τινησίας για το νέο σύνταγμα και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για την Αραβική Άνοιξη να έχουμε μία χώρα με ένα σύνταγμα και μάλιστα κατάφερε την Ισία να ολοκληρώσει το δικό της σύνταγμα πριν ολοκληρώσει η Τουρκία τις αντίστοιχες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Τουρκία, θα ήθελα να πω ότι ο Επίτροπος Φίλε έστειλε ε, τρεις επιστολές στην τουρκική κυβέρνηση. Μάλιστα δημοσιεύθηκαν και στον τύπο οι επιστολές αυτές. Η δική μας αξιολόγηση για τις μεταρρυθμίσεις ε, στο δικαστικό κλάδο και στο Ανώτατο Συμβούλιο ε, των Δικαστών. Ε, η αξιολόγηση μας λοιπόν δείχνει ότι όντως υπάρχει δρόμη σε σχέση με την προηγούμενη μεταρρύθμιση γιατί θέτοντας το δικαστικό κλάδο υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουμε παραβίαση της διάκρισης εξουσιών και παραβίαση του κράτους δικαίου. Εμποδίζεται η ανεξαρτησία, η αμεροληψία και η αυτονομία των δικαστών. Τελικά ελήφθη απόφαση για διακοπή της διαδικασίας έγκρισης αυτού του νομοσχεδίου και δεν αποσύρθηκε το σχέδιο αυτό προς το παρόν από συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως ε, έχει σαφή εντολή για την διαπραγμάτευση με την Τουρκία και την παρακολούθηση των δικαστικών μεταρρυθμίσεων. Θα ασκήσουμε στο έπακρο το περιεχόμενο της εντολής μας. Επίσης, ζητήσαμε διευκρινήσεις ε, για την πορεία της μεταρρύθμισης αυτής, για το κατά πόσο το νομοσχέδιο αυτό θα αποσυρθεί μερικός ή ολικός ζητήσαμε διευκρινήσεις και αν να γίνει πλήρης ανάκληση υπό ποιους όρους. Εμείς ε, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ε, για την Τουρκία για το κεφάλαιο 23, γιατί το άνοιγμα στις διαπραγματεύσεις του κεφαλαίου 23 θα είναι το καλύτερο σε ό,τι φορά τη δικαστική συνεργασία. Ε, μη θα ενισχύσουμε τις εργασίες μας με την ε, Τουρκία για να επεξεργαστούμε τα θέματα του κεφαλαίου 23. Πάντως θέλουμε η Τουρκία ε, να ε, σεβαστεί το κράτος δικαίου στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραγωνιστεί το κράτος δικαίου, γιατί καμία δημοκρατία δεν βρίσκεται υπεράνω του δικαίου. Πάντως μετά από πολύχρονες μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, μετά από δεκαετίες μεταρρυθμίσεις, έχουμε αισιοδοξία και πιστεύουμε ότι θα είναι ανθεκτικές και εύρωστες οι ε, κρατικές δομές της ε, Τουρκίας και θα αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Γιατί οι αστυνομικές και αντιδικαστικές αυτές ε, μεταρρυθμίσεις το τελευταίο καιρό ήταν κάπως ανησυχιστικές. Πάντως, υπό τον όρο ότι και η κυβέρνηση θα δείξει εμπιστοσύνη στις κρατικές δομές που δημιούργησε η ίδια, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αίσια έκβαση στην Τουρκία και η κυβέρνηση θα πρέπει να αφήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς να υλοποιήσουν το έργο τους και να μην υπονομεύει με την εισαγωγή αναδρομικής νομοθεσίας ε, τη διεξαγωγή του έργου και της αποστολής τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε παρακαλώ να απαντήσετε. Θέλω να πω μόνο ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας, ε, κυρία μου. Παρακολουθούμε και εμείς την κατάσταση στην Τουρκία πάρα πολύ προσεκτικά, από πολύ κοντά. Έχω κάνει και δήλωση για το νομοσχέδιο αυτό. επίσης ε, είπα και επανέλαβα και τη δήλωση του Πρόεδρου Γκιούλ την πρόσφατη ε, για το σεβασμό ε, των διεθνών προδιαγραφών και τη συμμόρφωση. Πρέπει να πω ότι λίγες μέρες πριν ο κύριος Γκιούλ είχε πει ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα δει και το συνταγματικό δικαστήριο. Σε περίπτωση λοιπόν που αυτό το νομοσχέδιο ακολουθεί στο δρόμο του, παρόλο που δεν το πιστεύω, γιατί προς το παρόν έχει διακοπεί, έχει ανασταλεί η διαδικασία, ε, θα αξιολογηθεί και από το τουρκικό συνταγματικό δικαστήριο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μποκίκιο. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας, να βοηθάτε όλους όσοι χρειάζονται τις συμβουλές σας ε, για την ε, οικοδόμηση θεσμών. Okay, friends, let's... Uh, λοιπόν, φίλοι μου, ας ε, συνεχίσουμε. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τις ιδιωτικές σας συζητήσεις, λυπάμαι πολύ. Ε. Αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε. Και συγκεκριμένα την κύρωση της συνθήκης για το εμπόριο όπλων, ο εισηγητής, ο κ. Αρνό Τανζό. Η κυρία Γκόμες γνωρίζω ότι θέλει να πει δύο λόγια πριν την ψηφοφορία, έτσι δεν είναι. Ναι, είστε σκιώδης συγγήτρια εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ναι, μάλιστα είμαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το έργο του και πρέπει να πω ότι δεν είχα την ευκαιρία να συνεννοηθώ μαζί του για αυτό που θα σας πω, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσει. Έχω μια πρόταση να κάνω. Προφορική τροπολογία, όποτε γίνεται, προστίθεται και συγκεκριμένα μου στην παραγραφό 19 όπου απλώς θα ψηφίσουμε και όχι μόνο θα υιοθετήσουμε ε, τις ε, συμφωνία της ΣΥΝΤΑ, θέλω να αναφερθούμε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, για την εφαρμογή των συστάσεων ε, στη συνέχεια που θα δοθεί ε, στη συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Δεν είναι απλώς ένα θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σαφώς θέμα εξωτερικών υποθέσεων. Στα κράτη-μέλη μας αυτό το έχουν αναλάβει τα Υπουργεία Εξωτερικών, τα Υπουργεία Εθνικής Αμήνης και πολλές φορές ή καμιά φορά ε, και το Υπουργείο Εσωτερικών επιλαμβάνεται, όχι το οικονομίας ή του διεθνού εμπορίου. Λοιπόν, όποτε υπάρχει τέτοια αναφορά για την εφαρμογή, να μην αναφέρεται μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όποτε περιορίζεται σε αυτό να προστίθεται και η η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μάλιστα. Βλέπω να συμφωνεί ο Παρακαλώ, κύριος Δανζό. Ναι, ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως, Πρόεδρε, με την Άννα Γκόμες. Θα δούμε περίπτωση σε ποιο άρθρο προτείνεται αυτό. Ε, αυτό που ανέφερε η Άννα είναι πολύ λογικό να προσθέσουμε εκεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, βλέποντας και κάνοντας λοιπόν. Δεν έχω αντίρρηση. Καλώς. Λοιπόν, είστε έτοιμοι όλοι να ψηφίσουμε. Αρχίζουμε. Τροπολογία παριθμό 5. Ψηφί Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Σημείο 7. Ψήφι Π. Ε, συγγνώμη, τροπολογία. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς, αρχίζει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 8. Ψήφι π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παριθμόν 9. Ψήφι π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Περάσει. Εγκρίθηκε. Θα πάμε τότε στην τροπολόγια περιφώνων 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος και πάλι για τη 15. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Να ξαναρχίσουμε. Γιατί 15 επαναλαμβάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα 16 ψηφί υπέ κατά Απόχες. Εγκρίνεται. 17 Επέ. Κατά. Απόχες. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ αυτό. 17. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Εγκρίνεται. 18 ψηφιπε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά στο ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 20 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 21. 21 ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 27. Όχι, 23 ψήφι πέρ, Κατά. Αποχές. We'll check this one. Έλεγχος χρειάζεται εδώ. 23. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Ε, κάποιος κατέβασε περισσότερα κουκιά μάλλον. 24 υπέρ της 24 κατά εποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 27 ψηφίπε κατά αποχές εγκρίνεται 28 είπε, Κατά. Α το ελέγξουμε αυτό καλύτερα. 28. Ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Πέρας. 19-15. Με μεγαλύτερη διαφορά αυτή. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Η 32, 32, 32. Υπέρ. Πατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. We'll check. So 32. We check. Vote is open. Εγκρίνεται. Όχι, ας το ελέγξουμε. 32. Άρχεται η ψηφοφορία και τελειώνει. Εγκρίνεται όντως. 33. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπε, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 3π Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 37 π Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίντα J Επέ κατά άποχες ας την ελέγξουμε αυτή είναι η J αρχής ψηφοφορία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου πέρας γκρίνεται 38 ψηφέ. κατά αποχές Χρειάζεται έλεγχος νομίζω. 38. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ωραία. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήταν D. Τροπολογία. Μια την προφορική της κυρίας Γκόμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Ίντα, F, ψήφιπε, κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η 40. Ψήφιπε. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Στις αιτιολογικές σκέψεις πάμε τώρα. 6. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Και τώρα. Οι αιτιολογικέ αναφορέ. Citations. 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και η 4. Και τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο αρχίζει. Πέρας. Καλώς συγχαρητήρια κύριε Ντονζό. Καλό αποτέλεσμα πετύχαμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι θα φύγετε παρακαλώ να το κάνετε αθόρυβα γιατί οι υπόλοιποι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Please. Please, the colleagues who would like to continue the discussion. Παρακαλώ, αφήστε τους συναδέλφους που θέλουν να συνεχίσουν τις συζητήσεις. Ε, αν έχουν ιδιωτικές συζητήσεις να κάνουν, το κάνουν εκτός αιθούσης. Γιατί θα περάσουμε στο θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση της κυρίας Γκόμες, έκθεση μάλλον της κυρίας Γκόμες, στην οποία και θα δώσω μέσα το λόγο. Άννα, σε ακούμε για τη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους τους και ηγητές με τους οποίους ε, έχω ήδη συναντηθεί και επεξεργαζόμαστε από κοινού κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες για να κερδίσουμε χρόνο συγχωνεύοντας κάποιες τροπολογίες. Θα ξανασυνεδριάσουμε και αύριο με τους και ηγητές, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για τις πολύ χρήσιμες και εύστοχες παρατηρήσεις τους. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση. Όχι γιατί Πρόκειται για την πρώτη φορά που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπονείται έκθεση για τη Σαουδική Αραβία, αλλά εξαιτία τη σημασία που έχει η Σαουδική Αραβία όχι μόνο στα θέματα σχέσεων με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για το ρόλο της ε, στην περιοχή και στον κόσμο γενικώ. Όπως είδαμε, επ' ευκαιρία της και στις συζητήσεις που κάνουμε με τους και ηγητές μπορούν να δοθούν διαφορετικές ερμηνείες για την πρόοδο των σχέσεών μας με τη Σαουδική Αραβία. Σίγουρα είναι σημαντική χώρα εταίρος από κάθε άποψη και το θέμα είναι να δούμε πόσο αποτελεσματικοί είμαστε εμείς στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας που είναι και κοινός μας στόχος άλλωστε. Πολλό μάλλον που οι αντιλήψεις για τη σημασία της προσάσπισης του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ίδιες, γιατί από πολλές απόψεις η Σαουδική Αραβία έχει διαφορετικές προσεγγίσεις από τις δικές μας για τα θέματα αυτά, για το θέμα των οικουμενικών αξιών και ούτω καθεξής. Άλλωστε, η Σαουδική Αραβία και νομικός δεσμεύεται από πολλές διεθνείς συνθήκες. Πάντως, εκτιμούμε την αλλαγή της δυναμικής που παρατηρείται στην Σαουδική Αραβία και σε αυτή την αλλαγή ο ρόλος των γυναικών είναι πολύ σημαντικός. Πολύ συχνά μιλούμε για τις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας εξετάζοντας μόνο ως θύματα και ως ανθρώπους, εξετάζουμε για τις περιπτώσεις ε, στέρησης των δικαιωμάτων τους. Αλλά διαπιστώνουμε ότι και ο ρόλος των γυναικών είναι θεμελιώδης στη Σαουδική Αραβία, γιατί δίνουν μάχη για την προάσπιση των ε, δικαιωμάτων τους, αλλά και για την αλλαγή σε ολόκληρη την κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας. Και μάλιστα το γεγονός ότι ε, έχουν τη δυνατότητα να μορφωθούν και να αποκτήσουν μεγάλες, πολλές γνώσεις και σημαντικά προσόντα και ακριβώς επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές θέσεις απασχόλησης ε, δίνουν μάχη και γι' αυτό, για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Γιατί από τη μια έχουμε τη Σαουδική Αραβία που είναι από τις σημαντικότερες, για να μην πω η, σημαντικ... η... η σημαντικότερη χώρα στον κόσμο, η χώρα με τις περισσότερους συνδρομητές Twitter. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό των ευκαιριών που δίνει το Twitter, αυτό το δίκτυο, για ανταλλαγή απόψεων. Μπορεί στην κοινωνία να μην έχουν τέτοια, τέτοιες δυνατότητες επαφής εξαιτίας ε, των κοινωνικών περιορισμών που ισχύουν και της ε, συντηρητικής ή πολύ σταλτικής ερμηνείας που δίνεται στις θρησκείες, αλλά εκμεταλλεύονται το Twitter για τις επαφές. Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις λοιπόν στην κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας, αλλά προσπαθούμε με επικοδομητικό πνεύμα να υιοθετήσουμε ένα πιο θετικό ρόλο στη Σαουδική Αραβία και δεν ε, αγνοούμε το σημαντικό ρόλο που παίζει η χώρα αυτή και στη σύγκρουση της Συρίας, για παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις στις σχέσεις ε, Σαουδικής Αραβίας ε, και Ιράν. και αυτές είναι εμφανείς ακόμη και εντός της Σαουδικής Αραβίας. Και πηγαίνοντας προάλλες στη Σαουδική Αραβία, λίγες μέρες πριν την σύναψη συμφωνίας για τη συμφωνία με το Ιράν, διαπίστωσα ότι υπήρχαν αρκετέ αντιστάσεις και επιφυλάξει ε, σε διάφορους κύκλους Σαουδική Αραβία. και μάλιστα έμεινα ευρώντητη διαβάζοντα ένα άρθρο που έλεγε ότι κάποιο μέλος βασιλικής οικογένειας δήλωσε ότι τώρα που η Δύση ε, θα καταλήξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της, ε, του Ιράν, τότε δεν έχουμε άλλη λύση παρά και εμείς να επαναφέρουμε το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Πακιστάν, το οποίο και χρηματοδοτήσουμε. Ε, χρηματοδοτήσαμε. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση. Και προσπάθησα να πείσω τους συνομιλητές μου στη Σαουδική Αραβία, παρόλο που ε, με διαβεβαίωσαν δεν είναι αυτή η κρατούσα γνώμη, υπάρχει παρόλα αυτά και αυτή η άποψη. Και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε μια τέτοια προσέγγιση να επικρατήσει. Κάτι άλλο που με εντυπωσίασε είναι ο τρόπος που κάποια μέλη, ακόμη και της ε, βασιλικής οικογένειας, αντιμετωπίζουν το κρίσιμο ζήτημα του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία και την διασπάθηση που γίνεται ταλέντων, γιατί δεν αξιοποιείται το τεράστιο ταλέντο που έχουν οι γυναίκες. Και φαίνεται ότι η χώρα έχει γίνει εχμάλωτος μιας μικρής ομάδας φονταμεταλιστών. Αυτό μάλιστα μας είπε και ο Υπουργός Πετρελαίου, που είναι και γιος ε, της, ε, ενός μέλους της πριγκίπισσας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Με ανησυχούν κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις. Έμαθα για παράδειγμα ότι κάποιοι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων φυλακίστηκαν και μάλιστα έχουν παραταθεί οι ποινές τους δεν θέλουμε φυσικά τέτοιες εξελίξεις. Εμείς άλλες εξελίξεις περιμένουμε από τις επαφές μας με τη Σαουδική Αραβία. Θα μπορούσα να μιλώ ετέρμονα, αλλά προτιμώ να σταματήσω για να ακούσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους που παρακολουθούν το θέμα. Και μια και η έκθεση δεν μιλά μόνο για τις σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και για το ρόλο της χώρας αυτή στην περιοχή, θα ήθελα να πω ότι ίσως ένα από τα πιο λεπτά σημεία και ευαίσθητα αφορά το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή. Πέραν του θέματος του Ιράν και της συγκρίσης στη Συρία που έχει γίνει ουσιαστικά έμεσος πόλεμος με συμμετοχή και της Σαουδικής Αραβίας και άλλων ομάδων που απέφχονται τις δημοκρατικές εξελίξεις στη ΣΥ. Αλλά θα προτιμούσα να ακούσω και τους συναδέλφους, γι' αυτό και θα διακόψω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάννα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι αυτή είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται για τη Σαουδική Αραβία η οποία έχει εξαιρετικό γεωπολιτικό και οικονομικό και γενικότερα πολιτικό ενδιαφέρον. Ε, γνωρίζουμε βέβαια ποια είναι η κατάσταση από πλευράς δικαιωμάτων σε σχέση με την υποστήριξη που κάνουμε εμείς στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα είναι η θέση των γυναικών, δηλαδή η ανδρική κυδαιμονία, η απαγόρευση να οδηγούν, ενώ σπουδάζουν οι γυναίκες εκεί και η μη αξιοποίησή τους ε, στις διάφορες θέσεις, πράγμα που θα μπορούσε να προσδώσει πολύ θετικό πρόσημο στη χώρα. Βέβαια γίνονται κάποια βήματα τελείως δειλά, όπως παραδείγματος χάρη τοποθέτηση των 30 γυναικών στην Σούρα, στην ε, Συμβουλευτική Συνέλευση, ή κάποιες ελπίδες που φαίνεται να διαγράφονται για τη συμμετοχή καταρχήν των γυναικών στις δημοτικές εκλογές με δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. Συμφωνώ με την κυρία Γκόμες ότι πράγματι η ισχυρή ομάδα είναι φονταμενταλιστές οι οποίοι και απαγορεύουν και την οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Και δεν μιλώ για χριστιανική θρησκεία ή άλλη, αλλά και τι μειονότητες στις Ισλαμικές. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, αλλά βέβαια η Σαουδική Αραβία είναι ένα σημαντικός παράγων για την ασφάλεια της περιοχής. Είναι γεγονός ότι συνεργάζεται με το δυτικό κόσμο ε, και βέβαια θα μπορούσε να συμβάλλει περισσότερο και ισχυρότερα στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής με ειρηνικά μέσα και στο ζήτημα της Συρίας ε, και στα υπόλοιπα ζητήματα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Ε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία και η χρήση βέβαια της ε, θρησκείας ως πολιτικού συστήματος είναι κάτι που κανέναν από εμά δεν βρίσκει σύμφωνος αλλά η, τα συμφέροντα της Ευρώπης όπως αντιλαμβάνεστε ε, λαμβάνουν υπόψη τους και την ισχυρή θέση που έχει η Σαουδική Αραβία στην περιοχή. Έχουν γίνει διάφορες τροπολογίες κύριε Πρόεδρε από διάφορες πλευρές. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση αρκετά επικοδομητική με την εισηγήτρια και ε, η δική μας πολιτική ομάδα ε, θέλει να τονίσει κάποιες θετικές ενέργειες που γίνονται και να ενθαρρύνει τη Σαουδική Αραβία να προχωρήσει περισσότερο. Δηλαδή θεωρούμε ότι η έκθεση δεν πρέπει να αποπνέει μια απόλυτα κατηγορηματική και αρνητική στάση ε, σε σχέση με το συγκεκριμένο κράτος και τις δυσκολίες που υπάρχουν για να μετατραπεί σε μια πραγματική δημοκρατία αλλά θα θέλαμε και η έκθεση να αποπνέει ενθάρρυνση ε, αυτών που ε, και ενδιαφέρονται να δουν τη χώρα τους διαφορετικά και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τις φωνές και τις αντιλήψεις τις πιο προοδευτικές μέσα στο χώρο. Αυτή είναι η γενικότερη γραμμή. Κατά τα άλλα θέλω να συγχαρώ την κυρία Γκόμες ε, για την έκθεσή της, ε, την οποία έκανε και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της επίσκεψης της εκεί επιτόπου και των συζητήσεων ε, που έκανε και νομίζω ότι και αύριο με τη συζήτηση που θα κάνουμε θα καταφέρουμε να βρούμε αρκετούς τελικούς συμβιβασμούς. Εμείς έχουμε εκφράσει την άποψή μας στην πρώτη συνάντηση ώστε να ψηφιστεί η έκθεση από την μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Νέιτ, ναι, τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Νάιτς. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκόμες και την πρωτοβουλία της να αναλάβει αυτή την έκθεση για τη Σαουδική Αραβία. Εκτιμώ ιδιαίτερως τις προσπάθειες τις οποίες έκανε για την προετοιμασία των συμβιβαστικών τροπολογιών που θα αντικατοπτρίζουν την μέγιστη δυνατή συνένεση. Όπως είπε και η κυρία Γιαννάκου, πιστεύω και εγώ, θα ήταν κάπως περίεργο η πρώτη έκθεση για τη Σαουδική Αραβία να περιλαμβάνει αποκλειστικά σημεία κριτικής. Αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να ξεκινήσει κάποιος διάλογος. Για να γίνει αυτό θα πρέπει φυσικά να υπογραμμίσουμε τις αξίες τις οποίες εμείς εμένουμε και ταυτόχρονα να δείξουμε, να αναγνωρίσουμε ότι διαπιστώνουμε τις αλλαγές οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό στη Σαουδική Αραβία και έτσι θα κρατήσουμε ανοιχτές τις διόδους επικοινωνίας με τους Σαουδάραβες. Είναι μια χώρα εξαιρετικά σημαντική, σε μια ιδιαίτερα ανήσυχη, θα έλεγα συνεχώς επικίνδυνη περιοχή. Η χώρα αυτή παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και έχει μεγάλη σημασία να παραμείνουμε σε καποφόρο επαφή, λέει η ομιλήτρια, με την Σαουδική Αραβία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι τους περνάει από το κεφάλι. Ούτε εμείς θα επικροτούμε τη χειροτέρευση της κατάστασης, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να πιέσουμε για μια σταδιακή αλλαγή και κάποιες θετικές σταδιακά εξελίξεις. Συγχαίρω λοιπόν και θα στηρίξω τις ε, ε, τροπολογίες, τις συμβιβαστικές της κυρίας ε, Γκόμες. Η κυρία Λόχμπίλερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα για μια καλή έκθεση και για πολύ συγκεκριμένες συμβιβαστικές προτάσεις, τις περισσότερες άλλωστε θα στηρίξουμε. Οι τροπολογίες μας σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σαουδική Αραβία προσωμιάζουν με τα προβλήματα τα οποία εντόπισε και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενέβης. Αναγνωρίζουμε κάποια βήματα προόδου, αναγνωρίζουμε όμως ότι δεν έχει υπάρξει συνολικότερα πρόοδος. Μια επιπλέον παρατήρηση εδώ. Είχα την χαρά να επισκεφθώ τη Σαουδική Αραβία και συζητήσαμε με τον Υπουργό Εσωτερικών τα θέματα αυτά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και ζητήσαμε στο μέλλον κάποιες δικαστικές διαδικασίες εναντίον εις βάρος αυτών που δραστηριοποιούνται στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα γίνονται ανοιχτά και θα παρακολουθούνται από τα μέσα ενημέρωσης και χαίρομαι που λέγω ότι έγινε ήδη αυτό σε μία περίπτωση, κάτι το οποίο με ικανοποιεί σε σχέση με τις δυνατότητες παρέμβασής μας. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν τις περισσότερες συμβιβαστικές τροπολογίες για την 7 σχετικά με τους μετανάστες. Εδώ θα θέλαμε να συστήσουμε να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με την διαδικασία σε εισαγωγικά σαουδοποίησης. Θα πρέπει επίσης να σας παραπέμψω και στην τροπολογία 28 την οποία εμείς είχαμε καταθέσει σχετικά με την διαδικασία αυτή. πως συνδέεται και με την καταπολέμηση της ανεργίας και με την κατάσταση των μεταναστών. Άννα θα ήθελες να κλείσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές σας παρεμβάσεις. Να σας ευχαριστήσω και για την συνεργασία που μου δείξατε για τις συμβιβαστικές. Πράγματι πρέπει εμείς να σταθούμε επικοδομητικά απέναντι στο θέμα Γνωρίζουμε ότι έχουν αναλυθεί αρκετές ε, πρωτοβουλίες και από τον βασιλέα της Σαουδικής Αραβίας και από την κυβέρνηση κάποια βήματα προώθησης ανθρωπιστικών ιδεών και συντήρησης ανοιχτής ε, του διαλόγου ε, για τις θρησκευτικέ ελευθερίες. Απ' την άλλη πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι η πραγματικότητα στη Σαουδική Αραβία μερικές φορές είναι διαφορετική. Ναι μεν από τη μία τρέχουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες για τον διάλογο προς τα έξω, απ' την άλλη εσωτερικά διαπιστώνουμε ότι δεν δέχονται κανένα άλλο δόγμα θα έλεγα με την εξαίρεση των ΣΥΙΤΟΝ σε ένα τμήμα της χώρας και δεν μπορεί η έκφραση της λατρείας να γίνεται δημόσια. Και αυτό σημαίνει ότι ε, εδώ αρνούνται τα θεμελιώδη θρησκευτικά δικαιώματα. Τώρα για, τους, για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι κάτι που μας προκαλεί ανησυχία και ευχαριστώ την κυρία Λόχμπίλερ για την επικοδομητική της στάση. Όταν είχα πάει στη Σαουδική Αραβία είδα ότι η διαδικασία σε εισαγωγικά σαουδοποίησης ήταν ένα βασικό βήμα το οποίο θα έδινε την δυνατότητα στην ένταξη ε, χιλιάδων παράνομων μεταναστών που δούλευαν ήδη εκεί και η διαδικασία αυτή δημιουργούσε κάποιες δυσκολίες ακόμα και ε, στις χώρες προέλευσης πολλών από αυτούς τους μετανάστες. Ξέρετε ότι 12 αεροπλάνα την ημέρα φεύγουν από τη Σαουδική Αραβία προς την Αιθιοπία με παράνομους μετανάστες και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό για μια χώρα σαν την Αιθιοπία και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν συνολικά διαφορετικά. Και μάλιστα έχουν υπάρξει και διώξεις, τραυματισμοί και θάνατοι. Ε, ακούσα για το θάνατο τριών Αιθιώπων ε, στα πλαίσια της δίωξής τους στη Σαουδική Αραβία. Ένας λοιπόν επιπλέον λόγος για να ε, πιέσουμε και να ζητήσουμε να υπάρξει δικαιοσύνη. Να υπογραμμίσω επίσης ότι θα λάβουμε υπόψη μας και την εξαιρετικά επικοδομητικές απόψεις της Επιτροπής Γυναικών του Κοινοβουλίου μας. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Βρισκόμαστε στην αρχή λοιπόν, είδαμε κάποια από τα προβλήματα, είδαμε επίσης ότι οι ομάδες συντονίζονται και η γνωμοδότηση θα καταλήξει θετικά. Έχουμε έξι λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη. Μια και δεν έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκράντι, ο οποίος είναι υπεύθυνο της Ούνρα για τους Παλαιστινίους στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει απλά να τον περιμένουμε. Θα ξεκινήσουμε σε 7 λεπτά.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 Ας ε, ξαναρχίσουμε. Έχει έρθει ο προσκεκλημένος μας, ο κύριος Φιλίππο Γκράντι, Γενικός Επίτροπος ε, του Γραφείου Αρρωγής και Έργων του ΙΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες στην Αγγής Ανατολή της Ούρα. Θέλουμε να τον καλωσορίσουμε ε, στην Επιτροπή μας. Είναι κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης εκτός από την εξωτερικών υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, Προσωπεί εδώ ο συνάδελφος Τέις ε, Μπέρμαν. Και όπως βλέπω από τα χαρτιά μου, η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ο κύριος Γκράντι ολοκληρώνει τη θητεία του στα τέλη Μαρτίου και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί αυτό και μια ευκαιρία για ένα γενικότερο απολογισμό και μια ανασκόπηση της θητείας σας με τα επιτεύγματα, τις δυσκολίες της και είμαι βέβαιος ότι τα ερωτήματά σας θα τον βοηθήσουν να μας κάνει αυτή την ε, ανασκόπηση. Όπως όλοι γνωρίζουμε δυστυχώς τα προβλήματα είναι όλο και πιο τραγικά εκεί για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες στη Συρία. Ως κοινοβούλιο Ανταποκριθήκαμε στα αιτήματα την Σούρα για επιπλέον υποστήριξη ήδη από την αρχή της σύραξης. Το πρόβλημα τώρα είναι θέμα δυνατοτήτων και βασικής υποστήριξης, ε, δηλαδή να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων εκεί. Μετά από αυτή την εισαγωγή θα παρακαλούσα τον συνάδελφο Τέις Μπέρμαν να πει δυο λόγια εξ ονόμα της Επιτροπής Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την Επιτροπή Ανάπτυξης αλλά και το γενικότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του με χαρά ακούμε πάντα τον Φιλίππο Γκράντι και τις αναλύσεις του. Σας καλωσορίζουμε. Ήμασταν στην Επιτροπή Ανάπτυξης ανέκαθεν κρυφνήσει υποστηριχτής ε, της ε, συνεχούς προσπάθειας ανακούφισης των δεινών που υφίστανται οι ε, Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Τώρα βρισκόμαστε στην τραγική συγκυρία που είστε υποχρεωμένοι να εργάζεστε εσύ υπέρ των Παλαιστινίων προσφύγων που είναι ξανά θύματα του εμφυλίου πολέμου στη Σύρια. Θα σας ακούσουμε, είμαστε πολύ περίεργοι να ακούσουμε την ανάλυση σας και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που είστε ακόμα σε θέση να επιτεχάνετε και θα θέλαμε επίσης να μας πείτε αν μπορείτε λίγο για την κατάσταση στη Γάζα και στα κατεχόμενα και στη Δυτική Όχθη, καθώς ε, συνεχίζει να συγκεντρώνει την προσοχή μας βεβαίως εκεί. Δεν θα μακρηγορήσω περαιτέρω, σας δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και σένα Ταΐς για τα καλά σου λόγια. Όπως είπατε, πιθανότατα θα είναι η τελευταία ενημέρωση που θα σας κάνω στην κοινή συνεδρία των επιτροπών. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω και διημών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και άλλα θεσμικά όργανα εδώ στις Βρυξέλλες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αντιπροσωπεία στην περιοχή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Η ΟΝΡΑ, πιστεύω και θα το εξηγήσω, παραμένει ένα σημαντικό θεσμό στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να μην είναι πάντα κεντρική και να κυριαρχεί στις συζητήσεις, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να παραγνωριστεί, πόσο μάλλον να αγνοηθεί. Έχουμε ε, ανάγκη την πολιτική υποστήριξη, την ηθική και την οικονομική και θα παραμείνει εκ των όνου κάνευ και το τονίζω αυτό για να έχουμε αποτελεσματική παρουσία. Μετά από 8,5 χρόνια στην Ούρα, λίγη η θητεία μου, την τελευταία τετραετία σχεδόν μέχρι σήμερα ε, διατέλεσα Γενικός Επίτροπος και σε δύο μήνες θα αποχωρήσω. Θα πρέπει να σας πω ότι συχνά ακούω ότι είναι δύσκολη καιρή για, για μένα και για τον οργανισμό μου, μου λέγουν. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι η ούρα είναι ένας ε, οργανισμός ε, ηλικίας 64 ετών που έχει συνηθίσει σε κρίσεις και έχει βοηθήσει ένα πληθυσμό που τώρα ενέρχεται σε 5 εκατομμύρια, είναι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες, ε, μετά από σύραξη, εκτοπισμό και επανειλημμένες και αποτυχημένες απόπειρες ειρήνευσης. Η παρούσα περίοδος μας δείχνει και πάλι ότι υπάρχουν κρίσεις και δυσκολίες συγκεντρωμένες, οι οποίες αλληλο επικαλύπτονται, συσσωρεύονται και κάνουν ακριβώς και πάλι τη ζωή των Παλαιστινίων προσφύγων ακόμα πιο δύσκολη. Πολλά είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν σήμερα την κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων και τη Σούρα. Θα ήθελα να αναφερθώ όσο μπορώ πιο σύντομα στα εξή. Πρώτον, ο πόλεμος στη Συρία και πώς επιδράσει τους Παλαιστινίου, Δεύτερον, η κατάσταση των Παλαιστινίων που ζουν υπό την Ισραηλινή κατοχή, αλλά ιδιαίτερα ε, ε, ο αποκλεισμός της Γάζας και ε, ο διχασμός στην ηγεσία των Παλαιστινίων. Τρίτον, η σχέση μεταξύ των ειρηνευτικών προσπαθειών και του θέματος των προσφύγων και το τέταρτο είναι ο ρόλος της ούρα και η πενιχρότηση των μέσων της. Θα σας αναφέρω μερικά πράγματα επιγραμματικά και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις στη συνέχεια. Για τη Συρία. 540.000 έχει μετρήσει η ΟΥΡΑ Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Συρία και μέχρι το 2011 και στις αρχές του πολέμου η ιστορία τους ήταν θετική. Δηλαδή, ανέκαθεν ε, την υποδοχή ε, υποδοχής και μεταχείρισης ε, θετικής στη Συρία με φιλοξενία. Ο πόλεμος είχε επίπτωση και σε αυτούς και από τις 540.000 πρόσφυγες πάνω από τους μισούς είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της Συρίας και επιπλέον ε, άλλες 80.000 ε, έχουν φύγει από τη Συρία για να γίνουν για δεύτερη φορά πρόσφυγες. Πώς επηρεάζει ο πόλεμος ε, την κοινότητα των προσφύγων και ιδιαίτερα των Παλαιστινίων. Είναι πολύ αντίστοιχος με τον τρόπο που βλέπουμε και σε άλλες κοινότητες. Ιδιαίτερα σε περιοχές που θεωρούνται στρατηγικές από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Γενικά βλέπει κανείς Κάποια στιγμή που ένοπλες ομάδες αντιπολίτευσης ελέγχουν κάποιες συνοικίες σε κάποιες πόλεις και θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, ε, προοδευτικά ε, ο Συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του περικυκλώνουν αυτές τις συνοικίες. Έτσι λοιπόν οι ε, άμαχοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές και προκειμένου οι Παλαιστίνοι που βρίσκονται παγιδευμένοι ταξίδια σταυρωμένων πυρών δεν μπορούν να ξεφύγουν ούτε να μπουν ούτε να βγουν από αυτή την περιοχή ούτε να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Αυτός είναι ο τρόπος που βλέπουμε να επηρεάζει τον άμαχο πληθυσμό πόλεμος και δεν εξαιρούνται οι Παλαιστίνοι από αυτό. Στο Γιαρμούκ, ξέρετε, δεν είναι καταβλισμός. Το Γιαρμούκ είναι προάστιο της Δαμασκού και μάλιστα εκτεταμένο όπου ε, διέμεναν περίπου 160.000 Παλαιστίνοι πριν φτάσει εκεί ο πόλεμος στο Γιαρμούκ. Είναι από τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Παλαιστινίων σε οποιοδήποτε μέρος εκτός Παλαιστίνης. Από το 2012 ο πόλεμος έχει φτάσει στο Γιαρμούκ λοιπόν ε, με αντιφρονούντες να ελέγχουν την πολύ στρατηγική αυτή συνοικία η προάστιο της Δαμασκού ε, και τους έχουν περικυκλώσει στη συνέχεια ο Συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του. 160.000 λοιπόν Παλαιστίνοι έχουν σχεδόν όλοι αποχωρήσει αλλά υπολογίζουμε 18 με 20.000 να είναι παγιδευμένοι στο Γιαρμούκ, παραμένουν εκεί. Και πρέπει να σας πω, από το Δεκέμβριο του 2012 ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας να φτάσουμε σε αυτούς. Πέρυσι και το καλοκαίρι καταφέραμε να τους στείλουμε κάποιο υλικό ε, προς ανακούφιση τους, αλλά από το Σεπτέμβριο και μετά τους τελευταίους 4-5 μήνες ήταν για μας απολύτως αδύνατο να κάνουμε οποιαδήποτε επιχείρηση στη Γιαρμούκ. Τα νέα που μπορεί να είδατε από τον τύπο είναι πάρα πολύ δραματικά. Ε, ο κόσμος λιμοκτονεί, σίγουρα υπάρχει υποσυτισμός ε, και ε, οι φέπουσες ασθένειες, δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, τα ανθρωπιστικά, τα οποία αναδύονται σε όλη την επικράτεια της Συρίας για κοινότητες που είναι απομονωμένες λόγω αυτού του πολέμου. Το τελευταίο διάστημα, 8 ημέρες ε, Μα ζητά επανελειμμένα η Συριακή κυβέρνηση να στείλουμε βοήθεια στο Γιαρμούκ. Μπορεί να το είδατε στον τύπο αυτό. Δύο απόπειρε ε, στέφσαμε επιτυχία περίπου. Αλλά για να σας πω πόσο αδύναμοι είμαστε. Μόνο 138 ε, δέματα στείλαμε. Ένα δέμα σημαίνει μια οκταμελή οικογένεια να καλύπτεται για 10 ημέρες. Άρα είναι σταγόνα στον ωκεανό για 18.000. Καταλαβαίνετε πόσο περιορισμένες είναι οι δυνατότητές μας. Και σας είπα, ε, πώς είναι η κατάσταση. Πηγαίνουμε ε, στα φυλάκια, μας λένε περιμένετε, περιμένουμε ώρες. Δύο φορές μας άφησαν να πάμε μέχρι τα σύνορα του Γιαρμού, την είσοδο, που ακόμα ελέγχει η Συριακή κυβέρνηση. Ο ε, κόσμος βγαίνει πολύ επιλεκτικά, με έλεγχο. Ε, ορισμένους δεν τους αφήνουν να πάρουν βοήθεια καν δεν τους επιτρέπουν. Μετά από ατέρμονες διαπραγματεύσεις ορών καταφέρνουμε να βοηθούμε μερικούς. Είναι πολύ ανισχυτικά αυτά που συμβαίνουν εκεί. Και θα ήθελα να κρώσω ένα κόδωνα κινδύνου. Μπορεί στο μέλλον αυτό να το ξαναδούμε, εάν και όταν επιτευχθούν κάποιες συμφωνίες για την ανθρωπιστική βοήθεια, που από ό,τι φαίνεται είναι το πρώτο βήμα των συνομιλιών της Γενέβης 2. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συμφωνηθούν αυτά στην κορυφή. Στη βάση θα αντιμετωπίσουμε αυτό. Εγώ δεν λέγω ότι θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο οι διαπραγματεύσεις αυτές να λάβουν χώρα γιατί είναι κατεπίγουσα η ανάγκη πρόσβαση για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Ας είμαστε όμως ρεαλιστές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμόζονται επί οι συμφωνίες αυτές. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προσπαθούμε να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο Γιαρμούκ και να διατηρούμε την πίεση προς όλες τις πλευρές. Όπως γνωρίζετε στη Συρία έχουμε 3.600 εργαζομένους, 10 θύματα δυστυχώς ε, είχαμε, ε, ε, σκοτώθηκαν και 20 αγνοούμενοι, δηλαδή είναι πολύ ψηλός ο φόρος αίματος που πληρώνουμε. Αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμαστε. Όπως Καθώς λοιπόν μας απασχολεί η Συρία δεν θα πρέπει να χάνουμε τη γενικότερη εικόνα. Τι σημαίνει αυτό για τους Παλαιστινίους. Είναι περιορισμένες οι δυνατότητές τους να αποχωρήσουν από τη χώρα. Γι' αυτό ε, ε, σας είπα ότι μόλις 80.000 εντό εισαγωγικών αποχωρούν. Οι περισσότεροι δεν τους επιτρέπεται να πάνε στην Ιορδανία αν πηγαίνουν στο Λίβανο. 51.000 τώρα έχουν πάει τουλάχιστον προσωρινά στο Λίβανο. Άλλο πρόβλημα και αυτό διότι γνωρίζετε ότι ο Λίβανος περίπου φιλοξενεί 250 ε, με 300 χιλιάδες Παλαιστινίους και τώρα εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως πάνω από ένα εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες. Η κατάσταση του Λιβάνου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και αυτοί οι 50 χιλιάδες Παλαιστίνοι δεν είναι τίποτα σε σχέση με τους Σύρους, αλλά πολιτικά και από όρους έτσι ευαισθησίας η παρουσία τους εκεί είναι πάρα πολύ ουσιαστική και πάρα πολύ κρίσιμη. Έρχεται λοιπόν να προσθεθεί δεν είναι μόνο ένα σύμπτωμα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία, αλλά και τι επίπτωση μπορεί να έχει γενικότερα στις όμορες χώρες. Γενικώ οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες θεωρούν ότι οι δυνατότητες που έχουν για μετακίνηση είναι πολύ πιο περιορισμένοι από ό,τι για τους Σύρους. Πήγα το περασμένο καλοκαίρι στη Συρία και μίλησα με Παλαιστίνιους πρόσφυγες που μου είπαν ότι τους θυμίζει η κατάσταση το 1948 όταν έφυγαν από την Παλαιστίνη. Το χειρότερο όμω είναι ότι τότε τουλάχιστον υπήρχε κάποια αλληλεγγύη και υποστήριξη, κάτι που δεν ισχύει πια στην περιοχή. Και αυτό λέει πολλά για την εξέλιξη της κατάστασης και την επιδείνωση της κατάστασης. Πάντως ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και χαίρομαι που το επισήμανε και ο κύριος Μπέργκμαν. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε όταν μιλούμε για τη Συρία την κατάσταση των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και στα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Δεν θα αναφερθώ εκτεταμένα στην Δυτική Όχθη, γιατί αυτό το συζητάτε συχνά. Στη Δυτική Όχθη ένα τρίτο του πληθυσμού είναι Παλαιστίνοι πρόσφυγες που υποφέρουν από τα ίδια δεινά από την κατοχή όπως και οι υπόλοιποι Παλαιστίνοι, κυρίως ε, εξαιτίας της αδυσόπιτης επέκτασης ε, των παράνομων ε, Ισραηλινών επικισμών. Θα επικεντρωθώ όμως στη Γάζα. Εκεί η αναλογία των Παλαιστινίων προσφύγων είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού, δύο τρίτα δηλαδή. Και εκεί φυσικά οι υπηρεσίες μας και το γραφείο μας ενεργοποιείται σημαντικά. Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες. Το 2010 το Ισραήλ αποφάσισε να ελαφρύνει κάπως ε, το, τον αποκλεισμό. Το χαιρετήσαμε αυτό και μπόρεσαν κάποιες ανθρωπιστικές οργανώσεις να ξεκινήσουν κάποιες, κάποια σχέδια ανοικοδόμηση. Αλλά πέρυσι είχαμε νέους περιορισμούς μετά την ανακάλυψη κάποιων σειράγκων και επίσης ε, άλλαξε η πολιτική της Αιγυπτιακής κυβέρνησης ε, γιατί έκλεισε όλα τα, τα σε ελαφρεμπορή και αυτό χτύπησε ανελαίητα τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας. Κανένας βέβαια δεν υπέρ των σειράγγων αυτών και του ελαφρεμπορίου. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την επιδίνωση που είχε σε ό,τι αφορά τη δρομολόγηση τη ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα τη Γάζα. ό,τι αφορά την εισαγωγή υλικών από το Ισραήλ, χρειάστηκε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία έκδοσης αδειών για την ενεργοποίηση κάποιων σχεδίων ανασυγκρότησης στη Λωρίδα της Γάζας. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε νέες εγκρίσεις αδειών. Πρόκειται για παλιά σχέδια που είχαν εγκριθεί, αλλά χρειάστηκε να επανυποβάλουμε αίτηση άδεια. Μόνο 12 όμως έχουν επανεγκριθεί μέχρι στιγμής και έχουμε 58 σχέδια ανασυγκρότησης ε, και νοικοδόμησης που περιμένουν ε, έγκριση από το Ισραήλ. Και μιλούμε μόνο για δικά μας σχέδια, τη Σούνρα, όχι για σχέδια και προγράμματα διμερών δωρητών. Πάνω από 100.000 ε, ευρώ σχέδια, 100 εκατομμύρια συγγνώμη, ευρώ ε, αξία σχέδια περιμένουν για έγκριση και είναι ελάχιστες ευκαιρίες που έχουν ε, οι άνθρωποι κάτι και της Γάζας για να απασχοληθούν. Έχουμε ελάχιστες βέβαια και μάλιστα τον Νοέμβριο του 2012 είχαμε κάποιες ελπίδες με την εκεχηρία και με την κατάβαση του πυρός, αλλά δυστυχώς ε, οι ελπίδες αυτές ε, εξανεμίζονται και δυστυχώς υπάρχουν ε, πιθανότητες για όλο και μεγαλύτερη κλιμάκωση και αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερω Γιατί μια νέα αναθέρμανση της σύγκρουσης στο, μετα στο της σύγκρουσης του Ισραηλοπαιστινιακού θα έχει οδυνηρές συνέπειες στη Γάζα και στην ειρηνευτική διαδικασία. Θυμάστε τι έγινε με την ε, προσπάθεια του 2009 και πώς επηρέασε την ε, ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Και μάλιστα οι περιορισμοί δυστυχώς οδήγησαν σε επιδείνωση των ανθρωπιστικών δικτών, ματέωση, δεινές οικονομικές συνθήκες, έξαρση της εκθετική άνοδος της φτώχειας, διάλυση των υποδομών. Αν δεν διαβάσατε τις περσινές εκθέσεις του ΟΗΕ για τη Γάζα με χρονικό ορίζοντα το 2020 θα δείτε τα τις προβλέψεις είναι τραγικές. Σας ε, συστήνω να τις εξετάσετε. Πριν τον αποκλεισμό θεωρούσαμε ότι ε, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η συλλογική τιμωρία, θα πρέπει, έπρεπε να έρθει ο αποκλεισμό και φυσικά θα αντιλαμβανόμαστε τις θεμητές ανησυχίες που έχουν για την ε, ασφάλεια το Ισραήλ και η Αίγυπτος, αλλά θα πρέπει αυτές να γίνονται εις βάρος της ανθρωπιστικής ασφάλειας στη Γάζα, το ενός εκατομμυρίου προσφύγων που βρίσκονται εκεί. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα να συνεχίσουν τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές ώστε να αποφευθεί μια νέα σύγκρουση και να προωθηθεί η συμφωνία για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός του 2000 12. Ελπίζω επίσης η διεθνής κοινότητα να συμφωνήσει και να στηρίξει τις προσπάθειες επανασυμφιλίωσης της Παλαιστινιακής ηγεσίας, γιατί μια κατακαιρματισμένη ηγεσία αποβαίνει βάρος της σταθερότητας της περιοχής και είναι επιβλαβής για το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας, για να μην αναφερθούμε καν στην ευημερία του Παλαιστινιακού λαού. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σχολιάσω είναι η ειρηνευτική διαδικασία. Είναι γνωστά αυτά τα θέματα, δεν θα επεκταθώ λοιπόν, λίγα μόνο σημεία Ας μην ξεχνούμε ότι το θέμα των Παλαιστινίων προσφύγων είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν επιτάπητο στα πλαίσια της ειρηνευτικής διαδικασίας και η επίλυση αυτού του παλιού ζητήματος είναι ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών όπως και τα επιμέρους θέματα γενικώ της τελικής ρύθμισης για το καθεστώς, και για να ευοδοθούν οι όλες, όλες οι συμφωνίες και να εφαρμοστούν όλες οι πτυχές της ειρηνευτικής διαδικασίας θα πρέπει να γίνουν ε, δεκτές και να γίνουν κτήμα των, ε, των λαών και κυρίως των Παλαιστινίων προσφύγων στην προκειμένη περίπτωση. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί ξέρουμε ότι μαζί με τα Ιεροσόλυμα το θέμα των προσφύγων είναι το θέμα με τη μεγαλύτερη σημασία, έχει υπαρξιακή σημασία και αξία και γνωρίζουμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν διστάμενες απόψεις ε, για το τι λύση είναι κατάλληλη. Φυσικά δεν πρόκειται η δική μου οργάνωση, η UNRWA, να λάβει θέση για το ζήτημα αυτό. Πάντως μπορούμε να σας ενημερώσουμε ότι ήδη υπάρχει μεγάλη ανησυχία για εν μέσω των προσφύγων και αυξάνεται αυτή όσο πλησιάζουμε προς την κατάληξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Πάντως, αν συνεχιστεί σε μια μεταγενέστερη φάση η ειρηνευτική διαδικασία, όπως όλοι ευελπιστούμε, θα είναι σημαντικό οποιαδήποτε λύση για τους προσφύγους να τηρεί το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ιδιαίτερα το ψήφισμα 194 και επίσης να ληφθούν υπόψη οι επιθυμίες των Παλαιστινίων προσφύγων και να προηγηθεί διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες κοινότητες. Και αυτό κυρίως ε, είναι ευθύνη της Παλαιστινιακής ηγεσία. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες θα πρέπει να είναι ενεχόμενοι στις ε, μελλοντικές διαδικασίες, γιατί θα πρέπει να, οποιαδήποτε συμφωνία να την κάνουν κτήμα τους, να μην θεωρήσουν ότι τους επιβάλλεται άνωθεν. Για να μην δημιουργηθούν ομάδες που θα είναι εχθρικές προς την ειρήνη και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για να περάσουμε σε αυτή την ε, φάση, στην επόμενη φάση. Πάντως αυτή η φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας μπορεί να ε, ακολουθήσει δύο πορείες, μία επιτυχή ή μία ανεπιτυχή. Αν είναι επιτυχής η ειρηνευτική διαδικασία, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ούρα θα είναι απαραίτητη σε μία χρονοβόρα και περίπλοκη μεταβατική περίοδο. Αν δεν στεφθεί με επιτυχία θα πρέπει να αποφύγουμε την κόπωση των δωρητών και να μην χαλαρώσει η στήριξη ή να αποσυρθεί η βοήθεια από τους Παλαιστινίους σε περίπτωση που δεν ευοδοθεί η ειρηνευτική διαδικασία και να αποσυρθεί και η βοήθεια, η στήριξη της ΟΝΡΑ. Αυτό θα είναι ακόμη πολύ πιο αρνητικό, θα επιτείνει την αποτυχία της διαδικασίας. Είναι σημαντική λοιπόν να μείνει αδιάλειπτη η υποστήριξη σας προς την Ούρα. Ξέρετε ότι έχουμε ε, προαιρετικές ε, ε, συνδρομές και παροχές. Παρόλο που ακριβώς επειδή προσφέρουμε κοινοφελείς υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προβλέψιμη η πόρη μας γιατί βοηθούμε σε νοσοκομεία, στην παιδεία, τέτοιου είδου υπηρεσίες δεν μπορεί να είναι απρόβλεπτες και δυστυχώς αυτό υπάρχει γιατί εξαρτώμαστε από οικειοθελεί ε, ε, παροχές και χορηγίε. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να συνεχίσουν να παραμένουν στην πρώτο πρωτοκαθεδρία και να υποστηρίζουν την ούρδρα και θα ήθελα να δίνουν περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο ε, δίνονται και είναι σημαντικά για να υλοποιηθούν οι υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στην υγεία και στην εκπαίδευση. Επίσης έχουμε το μισό από τη βοήθεια αυτή που δίνεται σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης όπως ανασυγκρότηση κτηρίων, ε, ε, ανοικοδόμηση οικειών και ούτω Βέβαια κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση του του προπολογισμού μας από τους δωρητέ, Δυστυχώς ε, αυξανόμενε είναι και οι ανάγκες και δεν ανταποκρίνονται στην αύξηση των κονδυλίων μας. Βέβαια, όταν δημιουργούνται συγκρούσει και δεχόμαστε συμπληρωματικού πόρους, δυστυχώς ε, ε, επιτείνονται και οι συγκρούσεις και δυστυχώς ο ρυθμός των χορηγιών δεν παρακολουθεί τον αυξανόμενο ρυθμό των συγκρούσεων και των προβλημάτων. Τους επόμενους μήνες η UNRWA θα υπογράψει την επόμενη ε, χρηματοπιστωτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα για τη συμβολή του στην UNRWA και μάλιστα μας ε, την αχύρα βοηθεία σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και στα τέλη του 2013 προτείναμε τα 80 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ε, το ετήσιο μερίδιο της ε, Συμβολής Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ούρα να αυξηθεί έστω και λίγο προκειμένου να έχουμε λίγο περισσότερο, μεγαλύτερο προϋπολογισμό προς το τέλος του έτους και ευελπιστούμε ότι θα γίνει δεκτή αυτή η πρόταση. Θα ήθελα εν κατακλείδη να πω ότι έκανα μια σύντομη περιγραφή δεδομένη έλλειψη χρόνου, μερικές από τις προκλήσεις που δημιουργεί ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και η κατοχή της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, το αποκλεισμό στη Γάζα, ο κατακαιρματισμό στην Παλαιστινιακή ηγεσία, η μεταβατική περίοδο στην Αίγυπτο, που επίσης επηρεάζει την κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων στη Γάζα. Και τα είπα όλα αυτά γιατί φοβούμαι ότι αυτή η πολύπλευρη κρίση πραγματικά έχει κάμψει το ηθικό των Παλαιστινίων προσφύγων, οι οποίοι έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, αλλά για πόσο ακόμη ε, θα, θα δείχνουν αυτήν την ανθεκτικότητα, πριν υποκύψει αυτή η ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητά τους σε μία απογοήτευση και ματέωση. Και μάλιστα από την 3η Δεκεμβρίου έχει απεργεί το προσωπικό μας γιατί ζήτησε αύξηση των των αποδοχών. Αυτό όμω δεν γίνεται γιατί έχουμε ελάχιστου πόρους. Αυτό δείχνει πόσα προβλήματα συσσωρεύονται. Το προσωπικό μας ζήτησε αύξηση των μισθών, φαντάζομαι είναι το ίδιο αίτημα πολλών δημοσίων υπαλλήλων, αλλά μίλησε για το πράσινο Γερμούκ στη Συρία, στη Δαμασκό, για την ειρηνευτική διαδικασία, τον αποκλεισμό τη Γάζας. Έχουμε πολυεπίπεδες προκλήσει και μία διασταύρωση προβλημάτων σε μία όλο και αυξανόμενη ανησυχία και αυξανόμενο άγχος και ταυτόχρονη προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα πιο πρόσφορο περιβάλλον και καλύτερες συνθήκες για την ειρήνη. Όταν ανέλαβα ως Γενικός Επιτρόπος της Ούνερα το 2010, τον Ιανουάριο του 2010, θεώρησα ως προτεραιότητά μου να αναπτύξω την εταιρική, εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΥΡΑ και να δημιουργήσω το να μετατρέψω το στρατηγικό διάλογο σε μια ουσιαστική εταιρική σχέση και όχι μια απλή τυπική σχέση μεταξύ ενός δωρητή και μιας οργάνωσης που λαμβάνει τους πόρους. Και Χαίρομαι για το διάλογο που είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την υπατεκπρόσωπο, με τους αρμόδιους επιτρόπους, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με άλλους ηθήνοντες ε, πολιτικούς. Ε, ήταν πολύ αγαστή αυτή η συνεργασία και θα ήθελα εν κατακλείδη να συνεχίσω να κρατήσετε αδιάλειπτη τη βοήθειά σας και τη στήριξη προ προς την ώρα και μάλιστα πρωτοστάτηση σε αυτή την υποστήριξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα αυτή να συνεχιστεί και προς το διάδοχό μου που θα αναλάβει επικεφαλής αυτής της δύσκολης οργάνωσης. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρμαν θα πάρει το λόγο τώρα comes as listened to συνήθως, ακούσαμε μια ξεκάθαρη παρουσίαση από τον κύριο Γκράντι. Σας ευχαριστώ για την ενέργεια την οποία επιδεικνύεται εδώ και τόσο καιρό που εργάζεστε για την Ούνρα. Θα ήθελα να θέσω ορισμένες ερωτήσεις βέβαια για την προϋπηρεσία σας τα τελευταία 8,5 χρόνια. Θα ήθελα να αξιολογήσετε λίγο τις, τα βασικά μαθήματα στα οποία πήραμε όλοι, αλλά να πω ότι μόλις έγινε μια έκθεση από, την, από το ελεγκτικό συνέδριο που ασκεί κριτική στον τρόπο χρηματοδότησης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μισθών χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων στη Γάζα που βρίσκονται σε υποχρεωτική ανεργία γιατί δεν τους επιτρέπει η Χαμάς να εργαστεί. Στον δημοσιονομικό έλεγχο λέγουν στην Επιτροπή την Κοινοβουλευτική ότι αυτά δεν τους αρέσουν και ότι πρέπει να σταματήσουμε τέτοιες γελίες καταστάσεις. Θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Άποψη δική μου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι για να διατηρηθεί η ζωντανή προοπτική μιας λύσης με δύο κράτη, θα πρέπει να συνεχίσει η πληρωμή προς τους δημοσίους υπαλλήλους της Παλαιστινιακής Αρχής όχι μόνο για λόγους ανθρωπιστικούς αλλά και πολιτικούς. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ειδική ερώτηση. Γενικά τώρα για τη Συρία και ιδιαίτερα για την κατάσταση στο Κόμς. Έχετε κάποια νέα ε, για την κατάσταση στην πόλη του Κόμς. Ε, πώς εμπλέκεστε εσείς σαν ούνρα. Η κυρία Γκόμες έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πράγματι η παρουσίασή σας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εσείς και η οργάνωσή σας κάνετε εξαιρετική δουλειά που δεν εκτιμάτε όσο πρέπει από τους πολίτες μας. Όχι από αυτούς που γνωρίζουν την ούνα, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου δεν συνειδητοποιεί την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνετε εξ ονόματος της διεθνούς κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση σωστά υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. Είναι και τεράστιες βέβαια οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζεται και οι οποίες από ό,τι φαίνεται ε, δυσκολεύουν όλο και περισσότερο, χειροτερεύουν όλο και περισσότερο. Να μας πείτε τώρα πια πώς βρίσκεται η κατάσταση στο, στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βήματα προς τη συμφιλίωση, δεν ξέρω αν πράγματι υπάρχουν. Άκουσα ότι υπάρχουν κάποια ενδιαφέρουσες προοπτικές. Αλλά ιδιαίτερα και μετά από αυτά που συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο άκουσα ότι άρχισαν να συζητάνε την πιθανότητα μιας συμφωνίας, μια συζήτηση που έγινε για εσωτερικούς περισσότερο λόγους, μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και κάποια τμήματα της ε, καφεστικίας τάξης ε, της Αιγύπτου ότι θα μετακινηθούν πληθυσμοί στην Χερσόνησο του Σινά και ότι αυτό θα λειτουργήσει σαν εγγύηση ε, για το ίδιο το Ισραήλ και για την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζα. Έχετε κάτι να σχολιάσετε γύρω από αυτό. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε κύριε Γκράντι, μπορείτε να απαντήσετε. για την ερώτηση την οποία έθεσε ο κύριος Μπέρμαν για τους δημοσίους υπαλλήλους της Παλαιστινιακής Αρχής που βρίσκονται αποκλεισμένοι στη Γάζα. Δεν μπορώ εγώ να μεταφέρω την άποψη της Παλαιστινιακής Αρχής γι' αυτό. Πάντως, οι σκέψει μου θα, ίσως θα πηγαίνουν λίγο πέραν της ερώτησής σας να πούμε γιατί έγινε αυτή η κατάσταση. Κάποιοι πληρώνονται και δεν εργάζονται. Γιατί. Γιατί υπάρχει αυτό το ρήγμα στην Παλαιστινιακή αρχή και γι' αυτό πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το ρήγμα. Εκτιμώ βέβαια ότι υπάρχουν πολιτικά κριτήρια πάρα πολύ ευαίσθητα τα οποία θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο ε, αντιμετώπισης. Εκτιμώ το ότι το κουαρτέτο έχει θέσει ορισμένους όρους που δεν έχουν εκπληρωθεί και οι διάφοροι τρόποι για την πιθανή επίλυση ε, των προβλημάτων αυτών και του ρήγματος ε, αν δεν υπάρξει τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το τι ε, θα μπορούσε κανείς να απαντήσει στην ερώτησή σας. Προφανώς και έχει σημασία να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ε, τον δημόσιο τομέα των Παλαιστινίων και τη Σούνρα και εμείς εξυπηρετούμε δύο διαφορετικά τμήματα του Παλαιστινιακού πληθυσμού, το λέω λίγο προκλητικά. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τη στήριξη και των δύο. Αλλά η δυσκολία αυτή ειδικά δεν αφορά μόνο την Ούνρα, αφορά την αρχή την Παλαιστινιακή και δεν θα υπάρξει λύση σύντομα. Και έρχομαι εδώ στην ερώτηση της κυρίας Γκόμες. Ξέρετε ότι διάφορες φήμες που ακούμε για μια κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφιλίωση. Αυτές οι φήμες που ακούτε εσείς τις ακούμε και εμείς, ότι τώρα όπου να είναι θα υπάρξει συμφωνία, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και από τις δύο πλευρές οι τελευταίες φήμες που ακούμε και με πολύ δυνατό τρόπο είναι ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Όταν το δούμε θα το πιστέψουμε. In terms, you know, I don't know about this transfer of people. I think that they seem to be a little bit as, you know, I may be wrong, but conspiracy theories. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες, σε πάση περιπτώσει, συνομωτικές οι οποίες ακούγονται. Αυτή τη στιγμή βέβαια η Αίγυπτος έχει να αντιμετωπίσει τα δικά της πάρα πολύ δύσκολα και περίπλοκα προβλήματα μετάβασης ανεξαρτήτως της λωρίδας. Πάντως εμείς και από τη δική μας πλευρά αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτό που βλέπουμε μάλλον είναι ότι η Αίγυπτος ε, ε, σκλήρινε τις σχέσεις της με τη Λωρίδα της Γάζας, ε, έκλεισε τα τούνελ τα οποία παρανόμως επέτρεπαν τη μεταφορά προϊόντων, αλλά θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι ο πληθυσμός της Γάζα, οι άμαχοι αν θέλετε, έχασαν έναν τρόπο προμήθειας αγαθών, καυσίμων, και άλλων ε, σημαντικών ε, υλικών για την καθημερινότητά τους και την επιβίασή τους. Είναι καλό λοιπόν το ότι δεν υπάρχει αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Αλλά δυστυχώς πώς θα περάσουν τα προϊόντα στα πλαίσια ενός εμπορικού αποκλεισμού πολύ αυστηρού. Αυτό είναι το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Για το HOMS εμείς δεν εμπλεκόμεθα άμεσα γιατί η συγκεκριμένη συμφωνία, αν κατάλαβα καλά, η οποία συζητήθηκε και στη Γενέβη, αναφέρεται στην παλαιά πόλη του Χόμς και στους αμάχους, που δεν είναι Παλαιστίνοι. Υπάρχει μια γειτονιά, ένα στρατόπεδο, ένα οικισμός παλαιστινιακός γύρω από την περιοχή αυτή, αλλά η περιοχή των Παλαιστινίων που κατοικείται από Παλαιστινίους και που επισκέφθηκα ελέγχεται από την κυβέρνηση οπότε δεν υπάρχει θέμα πρόσβαση στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή προς το παρόν. Αλλά η εξέλιξη αυτή είναι καλή γενικότερα. Ελπίζουμε εμείς ότι εάν οι διαπραγματεύσεις γύρω από την πρόσβαση στο Χόμς ε, ε, στεφθούν από επιτυχία θα ε, οδηγήσει σε αντίστοιχες λύσεις και για το Γιαρμούλκο όπως σας είπα προηγουμένως. Θέλετε να σας πω και άλλα. Τι άλλο να πω. Για τα διδάγματα που μπορεί κανείς να εξαγάγει. Να σας πω το εξής. Is that Το σημαντικότερο είναι ότι ε, στην οκταετή μου θητεία στην ώρα παρατήρησα το εξής η διεθνής προσοχή και υποστήριξη και ιδιαίτερη επιπλέον υποστήριξη ερχόταν πάντα σε περίοδους κρίσης. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στην επιχείρηση Cast το 2008, το Δεκέμβριο και το Γενάρη του 2009. Ήταν πολύ μεγάλη υποστήριξη ε, για τη δουλειά μας και για τους αμάχους που εκατέρωθεν πλήττονται. Ήταν κατακλειστική η υποστήριξη. Ε, αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι είναι πιο δύσκολο, διότι δεν είναι στο κέντρο της σύγκρουσης η Παλαιστίνη, έχουμε αποτελέσματα για τις επίγουσες δράσεις μας στη Συρία, διότι είναι κρίση και κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν υπάρχει η οξία κρίση ή τεράστια ορατή κάθε στιγμή. Και εκεί είναι η δυσκολία να επιτύχει κανείς πόρους. Αλλά όταν δεν μας δίνονται εμάς ε, χρήματα, και σε εμάς και σε άλλους όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γάζα, αυτό συνεισφέρει για την εκδήλωση της κρίσης και όταν ξεσπάσει η κρίση είναι αργά. Δηλαδή δεν δίνεται αρκετή προσοχή στις παραμονές μιας κρίσης και μπορεί η Λωρίδα της Γάζας αυτή τη στιγμή να ζει μια τέτοια φάση. Μετά είναι τεράστια ε, η ευθύνη και κοστίζει και πολύ περισσότερο. Βασικό δίδαγμα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε πολύ νωρίτερα, το είπε και η κυρία Γκόμες, και να γνωστοποιούμε στο ευρύ κοινό τι κάνουμε, όχι μόνο εμεί, αλλά και η δική μα οργάνωση, γιατί είναι απολύτω απαραίτητη αυτή η βοήθεια. Δεν είναι η μοναδική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και συνεισφέρει στη σταθερότητα της περιοχής που χρειάζεται κατεπηγόντω και τεράστια η ανάγκη αυτή τη υποστήριξη. Παρακαλώ να μην χαλαρώσετε τη δική σα υποστήριξη. Εμεί δεν θα λύσουμε τα προβλήματα, ούτε είναι αυτό ο σκοπό μα, αλλά μπορούμε να αποφύγουμε χειρότερε κρίσει που όταν θα ξεσπάσουν ε, θα σημαίνουν και πολύ μεγάλο κόστο γενικότερα και οικονομικό. Ο κύριο Μπέρμαν, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω γι' αυτό και να πούμε πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα για το Λίβανο. Είναι τεράστιος ο πληθυσμός τώρα των σύρων προσφύγων και πιέζει πάρα πολύ ε, και ε, τη χώρα και είναι και σημαντικό βάρος. Αυτό τι σημαίνει τώρα για την ούρα. Και είναι αυτή μια κλασική κατάσταση όπου λέτε εσείς καλύτερα να προλάβουμε τώρα παρά να τρέχουμε να θεραπεύσουμε μετά. Ναι, έχετε δίκιο. Τι σημαίνει αυτό για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες. Για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο. Οποιαδήποτε κλιμάκωση στο Λίβανο εσωτερικών εντάσεων που θα υποδαβλίζεται έξωθεν ή και όχι, ε, ε, θέτει σε κίνδυνο τους Παλαιστινίους που ήταν 300.000 συν 50.000 τώρα. Σε πολλούς κινδύνους. Παραδοσιακά ήταν ένα ευαίσθητο στοιχείο οποιασδήποτε εσωτερική σύγκρουση στο Λίβανο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ο πρόεδρος Σαμπάς, η ηγεσία των Παλαιστινίων στο Λίβανο και η Λιβανική κυβέρνηση την τελευταία δεκαετία είχαν πολύ καλή ε, δράση ε, για να κρατήσουν όσο μπορούν περισσότερο τους Παλαιστινίους εκτός των εντάσεων. Αλλά δεν είναι και πολύ μακριά. Είναι τεράστιοι οι καταβλισμοί, φτωχοί, ε, γεμάτοι εντάσεις και οι ίδιοι, πάρα πολύ ασταθείς και με πολύ λίγους πόρους. Εάν αυτοί οι καταβλισμοί δεν υποστηριχθούν και το λίγο που μπορούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά χρειαζόμαστε χρήματα, τότε αυτός ο εύθραυστος χαρακτήρας και ο κίνδυνος να εμπλακούν σε ευρύτερε συγκρούσεις στο Λίβανο είναι πολύ μεγάλος. Και ξέρετε ότι πολύ ε, γρήγορα εκρήγνυνται οι καταστάσεις αυτές όπως είδαμε το 2008. Δίπλα είναι η Συρία με τόσες πολλές εντάσεις ε, να αντικατοπτρίζονται από εσωτερικές τάσεις στο Λίβανο. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος και μεγάλος ο κίνδυνος να συμπαρασυρθούν και οι Παλαιστίνοι με μεγάλες και ε, επικίνδυνες ε, εξελίξεις. Έχουν και πολλά όπλα στους καταβλισμούς οι Παλαιστίνοι. Η πρόληψη πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι πολιτική να υποστηριχθεί η Λιβανική κυβέρνηση και η πρόληψη θα ήταν αληθή ας πούμε η κρίση και η σύγκρουση στη Συρία. Αλλά δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό. Αλλά από πολύ μικρότερο πρίσμα να μας βοηθάτε εμά και αυτούς που εργάζονται στους καταβλισμούς, βελτιώνουμε τις υποδομές τους, δίνουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, προσπαθούμε να βρούμε κάποιες δουλειές. Μπορεί να είναι μικρή ε, η συνεισφορά μας, αλλά βοηθάει στη σταθερότητα και αυτό το λιθαράκι μας. Okay. Uh, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξηγήσει σας. Οι συνάδελφοι έμαθαν πολλά και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις τους και θα παρακαλούσα τον κύριο Μπέρμπαν να κλείσει. Ε, Φιλίππο, είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω από το Μάρτιο και μετά πού θα καταλήξεις. Ποια θα είναι η νέα σου θέση και τα καθήκοντα που θα αναλάβεις. η Επιτροπή Ανάπτυξη του Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονε για την προσπάθεια σου και μπορεί η ώρα να υπολογίζει στη συνεχή μα υποστήριξη για να βρούμε και να υποστηρίξουμε την επαρκή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ το δικό σου οργανισμό. Θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή παρόλο που γνωρίζουμε ότι Αν είναι ένα πράγμα που στον κόσμο που έχει προκαλέσει τέτοια ματέωση είναι το θέμα των Παλαιστινίων προσφύγων. Και έχω εκπλαγεί που έχεις ε, ε, επιβιώσει ε, με την καλή έννοια και με, μεταφορικά μέχρι τώρα, αλλά δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φέρετε ότι είχες, έχεις διατελέσει δημοσιογράφος εσύ σε προηγούμενη ιδιότητα. Όπως και εγώ καθηγητής άλλωστε, αυτά δεν κρύβονται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι έχουν γίνει φωτογραφίσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Εθνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον κύριο Μοχαμέντα Αχμέτ Αλμούρ, καθώς και τον κύριο Άλτο Μπαϊσί, τον αντιπρόεδρο του Ομοσπονδιακού Εθνικού Συμβουλίου και την κυρία Αντζέλικα Νίμπρε, που είναι η πρόεδρο τη Αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Αραβική Χερσόνησο. Επίση καλωσορίζουμε και τα υπόλοιπα μέλη τη Αντιπροσωπείας και να ευχαριστήσω θερμά του τους και να ευχηθώ ταχύ ανάρρωση στον, προ, στον εξοχότητο Λίφα, τον επικεφαλής αποστολής σας και όπως είπαμε αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για μια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Ομοσπονδιακού Εθνικού Συμβουλίου σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με τη δυνατότητα αυτή. Αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι το πρώτο βήμα ενός πολύ μακριού δρόμου, όπως λένε και οι Κινέζοι. και θα μιλήσουμε για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Γιατί οι σχέσεις μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι πολύ σημαντικές. Όχι μόνο για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι σημαντικές ιδιαίτερα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξοχότατε, έχετε το λόγο. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Νίμπλερ για την πρόσκληση. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς ε, και εγώ και οι συνάδελφοί μου που ερχόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για μας ε, τους ε, Άραβες και Μουσουλμάνους η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός θεσμός με νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και επίσης έχει πολύ σημαντική ιστορική εμπειρία. Όπως ξέρετε, πολύ, πολλές σημαντικές επιστημονικές ε, ανακαλύψεις και εφευρέσεις έγιναν στην Ευρώπη και πολλές ιδέες για τη διάκριση των εξουσιών, για παράδειγμα, μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής Όλες αυτές οι ιδέες αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη. Από το Βρετανικό κίνημα για το Σύνταγμα, από τη Γερμανική παράδοση και πέρασαν από τις ε, διάφορες φάσεις της ευρωπαϊκής ε, ιστορίας. Και όλη αυτή η ιστορία, η διαδικασία, πέρασε και στον αραβικό κόσμο εμπνευστήκαμε πολλά από την Ευρώπη και για τα πολιτικά μας συστήματα και για την διοίκησή μας και για τις διάφορες πτυχές της ζωής. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι καινούρια. Ξεκίνησε από το 19ο αιώνα όταν είχαμε την ε, τόμο τον Μοχάμεντ Άλλη, τον αντιβασιλέα της Αιγύπτου που πήγε να σπουδάσει στο Παρίσι. Βέβαια δεν ήταν πάντα ειρηνικές και ευτυχείς οι σχέσεις μας. Είχαμε κάποιες φάσεις βίας, κυριαρχίας, πολλών και διαφόρων προβλημάτων στις αμοιβαίες σχέσεις μας. Ε, ταυτόχρονα όμω ένα μεγάλο τμήμα της αραβική αραβικής ιντελιγέντσια ε, έμεναν έκθαμβοι και θαύμαζαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτό το βλέπετε σε διάφορα βιβλία, σε πολλά γραπτά και πολλά θεσμικά μας όργανα και πολλοί θεσμοί ε, δημιουργήθηκαν και θεσπίστηκαν κατά το ευρωπαϊκό μοντέλο. Στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, ε, πολλές νομοθεσίες ε, ακολούθησαν ευρωπαϊκά πρότυπα και συστήματα ανώτερης εκπαίδευσης επίση μιμήθηκαν ευρωπαϊκά συστήματα εκπαιδευτικά. Οπότε η Ευρώπη ήταν ανέκαθεν για μας πηγή έμπνευσης εξαιτία των διαφόρων επινοήσεων, ανακαλύψεων, ε, της ευρωπαϊκής σκέψης και της συνεισφοράς της ευρωπαϊκής σκέψης στον ανθρώπινο πολιτισμό και στην ανθρώπινη εμπειρία. Όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή ο αραβικός κόσμος διανύει πολύ ευαίσθητους καιρούς. Και διάβασα σε ένα εβδομαδιαίο αγγλικό περιοδικό, στο Spectator, ένα κύριο άρθρο που μίλησε για τον θρησκευτικό πόλεμο μεταξύ Συνητών και Σιητών και το συνέκρινε με τον Τριακονταετή πόλεμο στην Ευρώπη. Και μάλιστα με πολύ απεσιόδοξο τρόπο το άρθρο αυτό μιλούσε για τον νέο πόλεμο που θα ξεσπάσει τον αραβικό κόσμο μεταξύ Σιητών και σουνητών και θα χρειαστούμε μια άλλη συνθήκη της Βεσφαλίας για να καταλήξουμε σε συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Και η Ευρώπη πέρασε τέτοιες εμπειρίες σε διάφορους πολιτικούς, σε πολλές πολιτικές φάσεις. Έχουν διαφορές γλωσσικές, θρησκευτικές, εθνοτικές και μεταξύ διαφόρων και διαφόρων αιρέσεων. Και επίσης θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που χρειάστηκε 200 χρόνια για να διαφθετηθεί. Είχαμε, είχατε 100 χρόνια του διαφωτισμού, είχατε 100 χρόνια επιστημονικών ανακαλύψεων, εφευρέσεων, σημαντικής έρευνας και την, επανάσταση, την βιομηχανική επανάσταση. Χρειάστηκε, χρειαστήκατε πολλά χρόνια στην Ευρώπη για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο και να αρμονίσετε τις διάφορες ιδέες, τις διάφορες θρησκείες, τις διάφορες αιρέσεις στην Ευρώπη. Και χρειαστήκατε πολύ χρόνο για την εξέλιξη των θεσμών σας και να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ιδεών, ομάδων. Ο αραβικός και ο ισλαμικός κόσμος δεν έχει περάσει από τις ίδιες ιστορικές εξελίξεις. Έχουμε ακόμη πολλά προβλήματα, έχουμε ακόμη πολλές ιδέες και οι διάφορες αραβικές χώρες πέρασαν από διαφορετικά στάδια εξέλιξης και ανάπτυξης και σε, σε πολιτικό επίπεδο, σε ε, πνευματικό επίπεδο. Και παρόλο που ένα μεγάλο τμήμα της κοινή γνώμης έχουν, τρέχουν μεγάλη συμπάθεια προς τις ιδέες του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις αξίες, τις οικουμενικές αξίες, ένα άλλο μεγάλο τμήμα της ε, κοινή γνώμης μας για πολλούς και διάφορους ε, λόγους δεν ξεχνά τις διάφορες ε, απικιακές βλέψεις, απικιοκρατικές βλέψεις, ακόμη και τα σχίσματα, τους θρησκευτικού πολέμους και τους θυμάται τους σταυροφόρους, τη και πολλά σημάδια στον αραβικό κόσμο και πολλοί κόσμος στον αραβικό κόσμο θυμάται όλες αυτές τις ε, φάσεις. Και ο αραβικός κόσμος με τους πολιτικούς μου στους θεσμούς και με το διαφορετικό ιστορικό θρησκευτικό υπόβαθρο και τις εμπειρίες σε σχέση με την απεικιοκρατία Μερικές φορές όταν αντιδρά σε μια κατάσταση στην Ευρώπη και βλέπει μερικές φορές πολύ αρνητική στάση της Ευρώπης απέναντι στο αραβικό κόσμο και φαίνεται ότι υπάρχει αμοιβαία παρεξήγηση για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον αραβικό κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν για να καταλήξουν συνεννόηση η Ευρώπη και ο Αραβικός και ο Ισλαμικός κόσμος ε, να γίνει εκτεταμένος διάλογος, πολλή συζήτηση. Και η κατάσταση δεν είναι μονόπλευρη. Δεν θα πρέπει η μία πλευρά να δίνει κηρύγματα στην άλλη για το ποια θεωρεί ότι είναι η καλύτερη λύση για τα διάφορα προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συνεχής διάλογος, όπως ξέρετε και στην πολιτική και στην οικονομία, αλλά και σε άλλους τομείς της ζωής δεν υπάρχουν στερεότυπες απαντήσεις. Γιατί η Ευρώπη δοκίμασε και τις, την, αγορά, την οικονομία της αγοράς, μετά πέρασε στην εθνικοποίηση, στην κρατικοποίηση, μετά στην ιδιωτικοποίηση. Τώρα προσπαθεί να, να δει το θέμα του επιχειρηματικού κύκλου. Είναι μια εξελικτική διαδικασία. Δεν υπάρχει ένα ιδεώδη σύστημα που να είναι κατάλληλο για όλους. Και έγινε και οι θεσμοί, έγινε διάφορα θεσμοί για να προστατευτούν διάφορες ομάδες κοινωνίας, για να έχουν όλη τη φωνή και εκπροσώπηση και την προστασία. Αλλά κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορική εξέλιξη και με διαφορετικό τρόπο οικοδόμησε τους θεσμούς της. Η Ινδία, για παράδειγμα, και η Κίνα έχουν κάθε μία το δικό της σύστημα. Και για να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα, της προκαταλήψεις, της παρεξηγήσεις και για να καταλήξουμε σε μία συνεννόηση, σε μία μηδέα κατανόηση, θα πρέπει να κρατήσουμε το διάλογο ζωντανό και συνεχή και να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το διάλογο δεν θα έχουμε αντιπαράθεση όπου ο καθένας θα διεκδικεί το δίκαιο του και θα προσπαθεί να βγάλει τον άλλο λάθος. Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Έχετε εσείς σταθερέ κοινωνίες, σταθερού θεσμού. Δυστυχώς ο αραβικός κόσμος δεν απολαμβάνει κάτι τέτοιο. Έχει σημαντικές ελλείψεις που τις είχατε κι εσείς στους παγκόσμιους πολέμους και στη μετάβαση από τα διάφορα συστήματά σας. Ξεπεράσετε τις αδυναμίες σας και έχετε φτάσει στην φάση αυτή σήμερα. Εμείς συνεχίζουμε τους πειραματισμούς, συνεχίζουμε αυτές τις διακυμάνσεις, προσπαθούμε να αναπτύξουμε τους διάφορους θεσμούς μας και δεν έχουμε μία ενιαία κοινωνία. Κάθε αραβική χώρα έχει τα δικά της προβλήματα και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Μερικές χώρες έχουν περισσότερο το θέμα των θρησκευτικών διαφορών με τις αιρέσεις. Σε άλλες χώρες έχουμε ε, φιλητικές διαφορές. Σε άλλες χώρες έχουμε διαφορά μεταξύ του στρατιωτικού, κατεστημένου και του πολιτικού. Δεν υπάρχει λοιπόν μία ενιαία λύση για όλο τον αραβικό κόσμο. Είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Και όπως ξέρετε, δυστυχώς, η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά την τελευταία διετία είχαμε κάποια θετικά δείγματα, κάποια αισιόδοξα δείγματα, που όμως στο μεταξύ έχουν δημιουργήσει μια βεβαιότητα και τώρα πια έχουμε πολλά αρνητικά σημάδια εξαιτίας του κόστου ζωή του βιωτικού επίπεδου, εξαιτία τη ε, μεγάλη φτώχεια, δολοφονιών. Είχατε κι εσεί τέτοια, έχετε γνώση για την κατάσταση αυτή, διαβάζετε καθημερινά εφημερίδε. τα βλέπετε στο διαδίκτυο, παρακολουθείτε τηλεόραση. Εμείς είμαστε ευτυχείς πάντως που είμαστε εδώ σε αυτό το σεβαστό διεθνές ε, οργανισμό Είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις μαζί σας, ίσως θα μην δώσουμε όλες τις απαντήσεις, αλλά είμαστε δεκτικοί και ελπίζω ο διάλογος να συνεχιστεί στο μέλλον. Δεν είναι μοναδική η συνάντησή μας εδώ σήμερα, θα σας συναντήσουμε και όταν έλθετε στη χώρα μας και σε διαφορετικά φόρα. Θα συναντηθούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συναντηθούμε επίσης και σε, σε, άλλες, σε άλλα συνέδρια για την επίλυση του προβλήματος της Συρίας, για τα θέματα του Αφγανιστάν. Γενικά έχουμε επαφές σε πάρα πολλά επίπεδα και προσπαθούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας και να συνεισφέρουμε και εμείς όσο μπορούμε έτσι ώστε να απαντήσουμε στα προβλήματα. Βέβαια είμαστε μικρή χώρα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε και να καλύψουμε όλες τις προκλήσεις του κόσμου, αλλά με τον δικό μας περιορισμένο τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επίλυση των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αναφερθήκατε στον 30 πόλεμο είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε εκεί που, που τέλειωσε μάλλον εκεί που είχε ξεκινήσει. Ξέρετε ότι Ρέγγιο, έγιους, ρελίγιο στα λατινικά. Ξέρετε ότι και ο Στάλιν είχε πει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα εγκατασταθεί η πολιτική εξουσία σε μία χώρα αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλής από τις στρατιωτικές δυνάμεις. Και εσείς έχετε περάσει από πολεμικές αναμετρήσεις και εμείς ε, ε, έχουμε περάσει από δύο πολέμους, ελπίζουμε να μην ε, συμβεί εκ νέου το ίδιο ποτέ πια. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται σε όλες τις χώρες όπως γνωρίζετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια εμπειρία την οποία συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες. Ε, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Νίμπλερ, ξέρετε ε, ότι τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα χρειάζονται πολύ μικρότεροι χρόνοι για να αλλάξουν ορισμένα πράγματα και γι' αυτό θα πρέπει μερικές φορές σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να ξεπεράσουμε τεράστιες δυσκολίες. Κυρία Νίμπλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξοχότατε. Ε, ε, εξοχότητε πρέσβοι, αξιότιμοι ε, καλεσμένοι. κύριε και κύριοι, αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα καταρχά να σα καλωσορίσω θερμότατα, εξοχότατε. Οργανωθείτε παρακαλώ λίγο με τα ακουστικά σας, γιατί μιλώ τη γερμανική. Παρακαλώ να βάλετε ακουστικά. Okay. Äh, Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, äh, äh, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εξ ονόματος της Αντιπροσωπείας για την Αραβική Χερσόνησο και να σας ευχαριστήσω κύριε Αλμούρ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή ε, αλλά και χαρά ε, η ευκαιρία που έχουμε σήμερα. Επισκέπτεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τους συναδέλφους σας. Σας καλωσορίζω θερμότατα και εγώ από πλευράς μου και θα ήθελα καταρχάς να σας πω και εγώ ότι ευχόμαστε στο ΣΕΙΧΙ καλήφα καλή ανάρρωση και ταχεία ανάρρωση και ε, να τον ξαναδούμε σύντομα υγιή. Παρακαλώ να του μεταφέρετε και να του διαβιβάσετε ε, τις ευχές μας. Η αντιπροσωπεία μας είχε τη χαρά και την τιμή να επισκεφτεί τη χώρα σας και το Ντουμπάι και το Αμπουντάβι είχαμε πολλές ε, επαφές και συνομιλίες και με εσά προσωπικά και με τους συναδέλφους σας και πρέπει να πω ότι και από πλευρά της δικής μας αντιπροσωπείας είναι σημαντικό να ανταλλάζουμε απόψεις. Το θεωρούμε πολύ χρήσιμο να προσπαθούμε να κατανοούμε ένα τον άλλον, να σεβόμαστε ένα τον άλλον. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές ε, θεωρήσεις, αξίες, ε, ιστορικές παραδόσεις και εξελίξεις και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος και εμείς στην Ευρώπη είναι γεγονός ότι έχουμε μακρά ιστορία, πολύ μακρά, πάνω από 200 έτη εμπειρίας ε, που συλλέξαμε για να καταλήξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη στον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης και δια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καθημερινά ακόμα αφιερωνόμαστε σε αυτές τις προσπάθειες. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ε, επαφές και ε, εμπειρίες με τις διαφορετικές παραδόσεις και ιστορίες στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αναζητούμε εκείνα που μας ενώνουν και να δούμε πώς από κοινού ε, μπορούμε και με τη δική σας ε, περιοχή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις χώρες ε, του Συμβουλίου του Κόλπου να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψη, να συνεργαζόμαστε και με την Ευρώπη και προς όφελος και των δικών σας πολιτών αλλά και των δικών μας. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο σεβασμό αλλά και θαυμασμό τις εξελίξεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ε, είπατε ότι σας εμπνέει η Ευρώπη, ισχύει όμως και το αντίστροφο και εμείς εμπνεόμεθα από τις δικές σας ε, εμπειρίες. Ε, είναι καταπληκτικό και μοναδικό το επίτευγμα που έχετε καταφέρει εσείς ε, στη χώρα σας και οι συνάδελφοι που είχαν μεταβεί εκεί στα Εμμυράτα έχουν ε, μείνει εντυπωσιασμένοι από αυτά που είδαμε. Πώς αναπτύσσεται το κράτος, πώς συμπαρασύρεται και ο πληθυσμός προς τον εκδημοκρατισμό. Είδαμε και πώς έχετε αναδείξει τις γυναίκες ε, που έχουν λάβει τη θέση τους και μεγάλες είναι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση. Όλα αυτά αξίζουν άκρατο θαυμασμό και αναγνώριση. Ε, ε, και η δική μας αντιπροσωπεία απέδιδε πάντα ε, πολύ μεγάλη σημασία στο να στείλουμε το μήνυμα ότι και στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ πιο στενά. Έχουμε το ευρωπαϊκό μας ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Mundus που γνωρίζετε ότι άνοιξε για να μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ε, από τις χώρες σας τα δικά μας πανεπιστήμια και το αντίστροφο. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, Φρονό, και χαίρομαι και ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία και πάλι από κοινού να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να συνεργαστούμε, ε, να έχουμε περισσότερη διασύνδεση. Και τελειώνοντας, Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δική σας ματιά και σκοπιά για την περιοχή σας. Πώς αξιολογείτε την κατάσταση, ας πούμε, στη Συρία. Ε, Ιδιαίτερα στα όσα συμβαίνουν και στο Ιράν που είναι κάποιες εξελίξεις που ε, αφορά η κατάσταση εκεί και τη γεωστρατηγική περιοχή και το Απουντάμπ και τα Εμμυράτα γενικότερα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρει πολύ να μάθει πώς αξιολογείται τα πράγματα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία, Πρόεδρε, να μιλήσω κι εγώ ως Πρόεδρος Αντιπροσωπείας και περιμένω με χαρά να ακούσω τις απόψεις σας από αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μιγιανμόν. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ στη μητρική μου γλώσσα. Ε, καταρχάς, να ενώσω και εγώ τη φωνή μου το καλώς ορίσατε προς τον πρόεδρο ε, Αλμούρ και την πολυάριθμη αντιπροσωπεία που σας συνοδεύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια για την Ευρώπη και ε, επίσης ελπίζω η επίσκεψη αυτή να συνεχιστεί από θετικά βήματα ε, περαιτέρω σύσφυξης ε, των σχέσεών μας με τα Εμμυράτα. Πρόσφατα προχωρήσαμε πάρα πολύ με την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίων για τους πολίτες των Αραβικών Εμμυράτων και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τούτον εκθέντο λοιπόν, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι οι διάφορες περιφέρειες του κόσμου ε, είναι πολύ διαφορετικές και ε, εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο. Είναι διαφορετικοί πολιτισμοί, οι κουλτούρες κτλ. Αλλά έχει δίκιο και ο πρόεδρος Πάσκου όταν αναφέρεται στην επιτάχυνση της ιστορίας. Η ιστορική χρόνη είναι διαφορετική σήμερα από 300 και 400 χρόνια πριν, το 17ο αιώνα. Οι Ευρωπαίοι ε, πραγματικά για ε, θρησκευτικούς πολέμους 30 χρόνια σκοτώναμε ένα τον άλλον αλλά ακόμα και στον 20ο αιώνα είχαμε δύο παγκοσμίους πολέμου. Ακριβώς γι' αυτό δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε ε, το ευρωπαϊκό έδαφος κάθε 30 χρόνια να ε, βάφεται στο αίμα. Βοήθησε πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ειρήνη, ε, για την ευημερία, για την οικονομική ανάπτυξη. Τώρα μας ενδιαφέρει να βγούμε από την κρίση και φαίνεται μακρινός ο πόλεμος. Εγώ εύχομαι στον αραβικό κόσμο ευημερία, ειρήνη, όλες τις δυνατές ελευθερίες για τους πολίτες, καλύτερη ολοκλήρωση, να μην υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών που είπατε ότι ε, αναφέρθηκε σε αυτή το περιοδικό Spectator. Ε, συμφωνώ και με την πρόεδρο Νίμπλερ, καλύτερο είναι να ακούμε εσά παρά ε, εγώ εμένα, γιατί γνωρίζω πολύ καλά τον εαυτό μου, αλλά θέλω να μάθω ότι πιστεύετε εσείς και πώς βλέπετε την ε, Αραβική Άνοιξη, τα όσα τεκταίνονται στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην Τινησία, πηγαίνουν καλά τα πράγματα, πώς το βλέπετε. Και αν μπορείτε να μας πείτε και τις προοπτικές σε σχέση με τη διάσκεψη Γενέβης 2 για τη Συρία και ε, την συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά ε, Παρακαλώ, αισθανθείτε εσά στο σπίτι σα και πείτε μας τι απόψει σα που είναι σημαντικές για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ το σεβαστό μέλος. Προσπάθησα να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα, γιατί όλοι σας έχετε παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις και στα μέσα ενημέρωσης και στα τηλεοπτικά κανάλια. Ξέρετε τι συμβαίνει. Πρέπει να κατανοήσουμε όμως τους μηχανισμούς που οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση. Όταν μιλάμε για τη Συρία, όπως ξέρετε, η Συρία και για 50 χρόνια είχε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ήταν πολύ αυταρχικό και το οποίο χρησιμοποίησε τον αραβικό εθνικισμό σαν κυρίαρχη ιδεολογία με, κάποιες, ε, με κάποια τμήματα επίσης σοσιαλισμού, εθνικισμού και λαϊκισμού. Στην ουσία απεδείχθη ότι ήταν ένα κόμμα ε, μίας οικογένειας, η οικογένεια Ασάντ με τον Μπεσίρελ Ασάντ και μετά με τον σημερινό πρόεδρο. Όταν ήρθε στην εξουσία ο Μπασάρ, υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε ένας διάλογος με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες έγινε αυτό που ονομάζαμε τότε η πολιτική άνοιξη της Δαμασκού αλλά πολύ γρήγορα το σύστημα έκλεισε όλες αυτές τις αιστείες συζητήσεων και επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση με ένα μόνο επιτρεπόμενο πολιτικό κόμμα και με μία οικογένεια, να μην πω με έναν άνθρωπο να ελέγχει το σύνολο της χώρας. Το σύστημα αυτό συνεχίστηκε για πολύ καιρό και οδήγησε αργότερα σε άλλες χώρες στο φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης, στην Τινησία, στην Αίγυπτο, στην Ιεμένη, τη Λιβύη και ακολούθησε η Συρία. Στην αρχή ήταν μια πολιτική κίνηση, ένα λαϊκό κίνημα αν θέλετε, όπου διάφορα τμήματα της κοινωνίας διαδήλωναν επιζητώντας ε, την ε, την κατάργηση του μονοκομματικού καθεστώτος και επιδιώκοντας την δημιουργία ενός πολυκομματικού συστήματος. Το κίνημα αυτό από την πρώτη στιγμή έγινε αντικείμενο καταστολής. Η καταστολή αυτή συνεχίστηκε για, μία περίπου ε, για ένα περίπου χρόνο. Υπήρξε λοιπόν καταπίεση, καταστολή, αλλά κάποια στιγμή κάποια τμήματα του στρατού βέβαια δημιούργησαν τον ελεύθερο Συριακό στρατό δημιουργήθηκε και μια πολιτική ηγεσία, η λεγόμενη συμμαχία πολιτικών ομάδων και κομμάτων και αυτά οδήγησαν σε μια ε, βίαιη ε, φάση. Υπήρξαν διάφορες ομάδες που στήριξαν τη σύραξη αυτή, ομάδες που προσπάθησαν κάποιοι να βοηθήσουν τους Σύρους ε, με διαφορετικές ιδιότητες η κάθε πλευρά. Στην αρχή υπήρξε προσπάθεια εξοπλισμού κάποιων ομάδων, το Ιράν, το Χεσμπολά, Ενεπλάκη και κάποιες άλλες χώρες πήραν μέρος στον εξοπλισμό των ομάδων και οδηγήθηκε στον εμφύλιο πόλεμο γιατί μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο όπως είχατε κάποτε στην Ισπανία εσείς. Ένας πάρα πολύ βίαιος πόλεμος αδελφοκτόνος πόλεμος. Η χώρα μας προσπάθησε να πάρει μέρος ε, στην κοινή προσπάθεια την οποία έκανε η διεθνής κοινότητα και σε περιφερειακό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δυστυχώς υπήρξε και ένα νέο στοιχείο το οποίο προσετέθη στην κατάσταση αυτή. Κάποιες ριζοσπαστικές α, ε, α, ε, ε, θρησκευτικές μουσουλμανικές ομάδες, η Αλνάσρα και μετά ο στρατός της Συρίας και του Λιβάνου ενεπλάκησαν. Όλα αυτά έκαναν την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη και οδήγησε και στη διαμόρφωση κάποιων απόψεων από τη μία η κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την άλλη η αντιπολίτευση η οποία είναι ιδιαιτέρως ακραία και όλα αυτά δημιούργησαν πάρα πολλές συγχύσεις. Στην αρχή τα πράγματα φαινόντουσαν απλά. Ο ελεύθερος στρατός με συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία με έδρα στην Κωνσταντινούπολη ή στην Αίγυπτο και αυτό προκάλεσε και τη συμπάθεια του υπολείπου κόσμου. Όταν ενεπλάγησαν τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Νάστρα και αυτός ο νέος στρατός της Συρίας και του Ιράκ και με αυτά τα οποία έκαναν εις βάρος των αμάχων άρχισαν να μοιάζουν με φασιστικές θρησκευτικέ ομάδες που ήθελαν να επιβάλλουν τη Σαρία. Και έτσι φτάσαμε στην κατάσταση αυτή. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Έχουμε πάρει στην προσπάθεια να χρηματοδοτήσουμε τα στρατόπεδα των προσφύγων στην Ιορδανία. Επίσης συμμετέχουμε σε προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών στα στρατόπεδα αυτά να μην χάσουν ε, τις δυνατότητες εκπαίδευσης τις οποίες ε, έχουν. Συνεργαζόμαστε με Ευρωπαίους φίλους στα πλαίσια της Γενέβης 1 και 2, ε, σε συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη, σε συναντήσεις στην, στην Ευρώπη, έτσι ώστε να κρατήσουμε ενιαία στάση. Υπάρχει ανάγκη να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά να πείσουμε την κυβέρνηση να μην ακολουθήσει ε, ε, την απαράδεκτη εγκληματική και δολοφονική τακτική που ακολούθησε μέχρι τώρα. Αν σταματήσουν να διαπράττουν τέτοιες ε, ενέργειες προφανώς και έχουν θέση στη νέα διακυβέρνηση της χώρας. Δεν γνωρίζουμε επίσης και ποιες ακριβώς μεγάλες δυνάμεις εμπλέκονται. Τι ακριβώς θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις. Θέλουν να επηρεάσουν απλά με πολιτικό τρόπο την κατάσταση. Ή μήπως κάποιες δυνάμεις ε, ε, πράγματι δεν θέλουν ε, η κυβέρνηση της χώρας αυτής να εκμεταλλεύεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες και θρησκευτικέ και φιλετικές και εθνοτικές. Ξέρουμε ότι οι Ρώσοι στηρίζουν το καθεστώς, αλλά μερικές φορές υπάρχουν αντιφάσεις στην πολιτική τους λένε σαν παράδειγμα ότι η μεταβατική νέα κυβέρνηση δεν θα περιλαμβάνει στελέχη της κυβέρνησης αυτής, μερικές φορές λένε το αντίθετο οι Ρώσοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια της Γενέβης, των συναντήσεων της Γενέβης εμείς όπως σας είπα υποστηρίζουμε πάρα πολλές ε, ανθρωπιστικές ενέργειες υπέρ της Συρίας. Έχουμε δώσει 200 εκατομμύρια δολάρια και για το νοσοκομείο το οποίο έχει 80 γιατρούς και νοσοκόμες ε, για να βοηθήσει στον τομέα της υγείας. Και θα συνεχίσουμε στην ίδια κατάσταση τους επόμενους μήνες. Ελπίζω να μην κρατήσει 30 χρόνια ο πόλεμος αυτός και να μην έχουμε και την καταστροφή του Λιβάνου όπου ο εμφύλιος πόλεμος κράτησε 18 χρόνια. και μόνο όταν συνήλθαν οι δύο πλευρές κατάφεραν να συμφωνήσουν σε νέο τρόπο διακυβέρνησης του Λιβάνου. Ξέρετε ότι όλες αυτές οι αλλαγές στην συμπεριφορά των Ρώσων συνάδουν με την πίεση έτσι ώστε η κυβέρνηση της Συρίας να υποχωρήσει σε διάφορους τομείς και σε άλλους όχι. Ο κύριος Αλαφράγκα, θα ήθελα και εγώ κύριε Πρόεδρε να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, τον Πρέσβη και όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα σας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής. Και ακούσατε τις ερωτήσεις για το ρόλο σας στην Αραβική Άνοιξη και ιδιαίτερα τις προσπάθειες που κάνετε για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την συνδρομή στους πρόσφυγες. Ξέρω ότι θεωρώ ότι στη ζωή, στην επιστήμη, στον πολιτισμό, την πολιτική και την κοινωνία το πιο σημαντικό για τους ανθρώπους είναι όχι μόνο να αναγνωρίζουν αλλά και να μπορούν να προσπαθούν να καταλάβουν, να κατανοήσουν. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική και καλό θα είναι να δώσουμε ε, να αναγνωρίσουμε όχι μόνο επιδεύματα της επιστήμης και της γνώσης αλλά και στον διάλογο, τον διαπροσωπικό και στην προσπάθεια αλληλοκατανόησης και σε αυτό το πλαίσιο του διαλόγου και της αλληλοκατανόησης θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί ακούσατε τις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση της αντιπολίτευσης ε, στην ε, χώρα σας. Πώς αντιμετωπίζει το Εθνικό Συμβούλιο την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς θα εμβαθύνεται μεταξύ των κομμάτων σε έναν επικοδομητικό και καρποφόρο διάλογο προκειμένου να ενισχύσουμε και να συσφίξουμε τους δεσμούς μας ως νομοθετικών οργάνων αλλά και τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση. Γιατί ξέρετε ότι εμείς έχουμε ε, προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού γιατί πρόκειται για οικουμενικά δικαιώματα. Θερμό καλωσόρισμα λοιπόν προς συναδέλφους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικό, ευαίσθητο και πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπους ε, για να έρθουμε πιο κοντά. Ευχαριστώ. Εξοχότατε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τμήμα των γενικών δικαιωμάτων των πολιτών και των υπηκών μιας χώρας, των κατοίκων μιας χώρας. Στις τελευταίες μας συναντήσεις ασχοληθήκαμε με μια πολύ σημαντική νομοθεσία που θα συμπληρώσει τις, τους υπόλοιπους νόμους που έχουμε και πρόκειται για τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι από ε, από Πρόκειται για μια πολύ σημαντική νομοθεσία και πραγματικά πρωτοπόρα στην ε, περιοχή της συνεργασίας του κόλπου, στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου μεταξύ των Αραβικών χωρών. Και φυσικά θεσπίσαμε πολλούς ε, νόμους. Μερικοί ανήκαν περισσότερο στην παλιότερη κοινωνία, αλλά εμείς είμαστε μια νέα χώρα και μια χώρα στην οποία ίσχυσαν κάποιες ε, παραδοσιακές αρχές, ε, ηθική, εθιμικό δίκαιο και στις σχέσεις μεταξύ των ε, ηγετών και των διαφόρων ομάδων της κοινωνίας. Ακόμη και σχέσεις γονέων και παιδιών. Τώρα στο μέτρο που μορφώνεται περισσότερο, εξελίσσεται περισσότερο και κλεπτίζεται περισσότερο η κοινωνία μας, αναδεικνύονται και νέα φαινόμενα. Και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινωνίας, οι σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών, μεταξύ των διαφόρων ομάδων της κοινωνίας, των, κοινωνικών τάξεων και οι σχέσεις με τους ε, εργαζόμενους μετανάστες, οι σχέσεις με τους επισκέπτες της χώρας μας αλλάζουν. Προσπαθούμε να μάθουμε από τους άλλους, προσπαθούμε να εξελιχθούμε. Και αυτή η διαδικασία είναι μια συνεχής διαδικασία. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και μερικές φορές προσπαθεί να παρακολουθήσει κάποιες άλλες εξελίξεις ή είναι ένα τμήμα της εξέλιξης μας της διοικητικής, της συνταγματικής, της ανέλυξης μας και από νομοθετική άποψη και της ορίμανσης μας όλους αυτούς τους τομείς. Πολλά πράγματα τα κάνουμε με βάση το παραδοσιακό μας σύστημα, με βάση τα παραδοσιακά πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Αλλά με, τη νέα, με, τη, με τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας θα θεσπίσουμε νέα νομοσχέδια θα θεσπίσουμε νέους κανόνες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Και όπως ξέρετε από διάφορες εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε μερικούς τομείς επωφεληθήκαμε από αυτή την εμπειρία. Στο παρελθόν ήμασταν μια πολύ απλή κοινωνία. Δεν είχαμε εμπόριο ανθρώπινων ανθρώπων γιατί δεν είχαμε καθόλου μετανάστες εργαζομένους. Ήταν μια κοινωνία με φυλές, δεν είχαμε καθόλου μετανάστες. Στο μέτρο που αρχίσαμε να εξελισσόμαστε και να υποδεχόμαστε και μετανάστες εργαζόμενους, διαπιστώσαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνονται θύματα εκμετάλλευσης, όχι από ντόπιου, αλλά και από άλλους αλλοδαπούς μερικές φορές που διαβίουν και εργάζονται στην πατρίδα μας, στις χώρες μας. Και αυτό μας οδήγησε στο να συστήσουμε νέες επιτροπές και θεσμούς στην κυβέρνηση για να μελετήσουμε αυτά τα φαινόμενα, να δούμε αν όντως πρόκειται για φαινόμενο ή αν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις γιατί θα πρέπει ανάλογα με τη διάγνωση κατάστασης να θεσπίσουμε κανόνες, να προβλέψουμε διαδικασίες για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προσαγάγουμε στα δικαστήρια αυτούς που ε, κακομεταχειρίζονται άλλους ανθρώπους, που τους εκμεταλλεύονται να τους διώξουμε ποινικά και ενδεχομένως να τους ε, τιμωρήσουμε και ποινικά. Έχουμε συγκροτήσει μία νέα επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάγεται στο Εθνικό μας Συμβούλιο. Αυτή η επιτροπή θα είναι μόνιμη. Δεν είναι μία ad hoc, μία προσωρινή επιτροπή. Αυτή η επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα εξετάζει τις νομοθετικές προτάσεις, τα διάφορα νομοσχέδια για να εξετάσει, να εξακριβώσει κατά πόσο ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πιο προηγμένων χωρών. Και θα συζητάμε την κυβέρνηση τα πιο περίπλοκα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, πολλές εκθέσεις αναφέρονται συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα των γυναικών. Πολλές φορές, διαβάζοντας τις εκθέσεις, έχουμε την εντύπωση ότι έχουν γραφτεί για άλλες χώρες, όχι για μας. Γιατί στη δική μας χώρα έχουμε γυναίκες υπουργού, γυναίκες ε, στη Βουλή, πρέσβυρες, διευθύντριες ε, σε σχολεία, εργαζόμενες και μάλιστα σημαντική, σημαντική στα πανεπιστήμια μας έχουμε γυναίκες σε πολύ κέρυες θέσεις. Και έχουμε επίσης παρουσία γυναικών σε όλα τα Υπουργεία, ακόμη και στο Υπουργείο Στρατού, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην αστυνομία έχουμε στελέχη γυναίκες. Επίσης, γυναίκες συμμετέχουν στο εμπόριο, έχουν δικές τους επιχειρήσεις οι γυναίκες ε, συμμετέχουν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν, όταν διαβάζουμε τέτοιες εκθέσεις, ότι έχουν γραφτεί για άλλη κοινωνία, όχι για τη δική μας. Γιατί δεν ισχύουν όλα αυτά για μας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν είμαστε τέλειοι από την άποψη αυτή. Και θα πρέπει σε πολλούς τομείς να σημειώσουμε πρόοδο, σε αρκετούς τομείς να εξελιχθούμε. Για παράδειγμα, για την αγορά εργασίας έχουμε δύο είδη μεταναστών, τους ε, ε, οικιακούς βοηθούς και τους εργαζόμενους σε εργοστάσια ή στον οικοδομικό κλάδο. Και την τελευταία δεκαετία όλοι οι εργαζόμενοι Τις οικοδομές, για παράδειγμα, έπρεπε να φοράν κράνη. Θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Θα πρέπει να μην δουλεύουν ε, όταν έχει καύσωνα. Και αν ε, υποβάλλονταν, αν είχαν παράπονα και προβλήματα με, την, ε, με τους εργοδότες τους, μπορούσαν να στραφούν είτε στα εργατοδικεία, για να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους, αλλά μπορούσαν να ε, υποβάλουν αγωγή και στα δικαστήρια, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Είχαμε και πολλές περιπτώσεις ε, για τους μισθούς. Και η κυβέρνηση επιμένει ο μισθός να πηγαίνει κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό των εργαζομένων, ώστε ο εργολάβος ή οποιοδήποτε εργοδότης τους απασχολεί να μην μπορεί να καθυστερήσει την καταβολή του μισθού. Γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση θα εντοπιστεί και θα καταγγελθεί. Υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν θέλω να πω σε πολλές μεγάλες λεπτομέρειες, γιατί οι συνάδελφοί σας μας επισκέφθησαν και αν έρθουν μελλοντικά σε άλλη επίσκεψη θα ε, τους δείξουμε τα διάφορα ε, αυτά θέματα και να μας κάνετε και παρατηρήσεις. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση, ε, βολή είμαστε. Εμείς μπορούμε να ε, συμβουλεύουμε την κυβέρνηση και να της θέτουμε υπόψη διάφορα θέματα. Έτσι έχει η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, εξοχότατε. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε 30 χρόνια στη διάθεσή μας, όπως κάποιοι άλλοι, για να κάνουν πολέμους σίγουρα αυτή η πρώτη επαφή ήταν πάρα πολύ καρποφόρα και νομίζω ότι γνωρίζετε ότι στο μέλλον θα αναπτύξουμε και άλλες σχέσεις και η συνάδελφος κυρία Νίμπλερ θα μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και την κυρία Αντιπρόεδρο, τη Δόκτωρ Κουράισι, καθώς επίσης και τον ε, πρέσβη, τον οποίο δεν αναγνώρισα προηγουμένως, τον πράττω τώρα όμως. Ε, καλωσορίσατε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε.